Not so easy. Good afternoon, everybody. Καλησπέρα Ελπίζω ότι θα έρθει κάποιο από το ΕΛΚ εδώ. Δεν ήρθε κανένα. Θα αρχίσουμε όλα αυτά εμεί τι εργασίε μα. Σημείο 8 τη ημερησία διάταξη. Κεφαλικέ απαιτήσει για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τι πράξει επαναιτητλοποίηση και ο επεπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών. Θα δώσω μέσα το λόγο στην εισηγήτρια Αρλίν Μακάρθη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σα κάνω μια γενική παρουσίαση, να ξεκινήσει η συζήτηση και μετά να σας ακούσω για να έχω απόψει και των σκιωδών και των συναδέλφων τη Επιτροπή που ενδιαφέρονται στο θέμα αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, νομίζω το υπόβαθρο είναι η χρηματοπιστωτική κρίση που είδαμε τις αδυναμίες ιδίως του τραπεζικού τομέα και οι συναδελφοί αναφέρονται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 2-3 εκατομμύρια ε, για την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα και η ομάδα των 20 σε διεθνές επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν ένα ευρύ πρόγραμμα α, μεταρρύθμισης για να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά διάφορες δυνατότητες όσον αφορά το φόρο παραδείγματος κάνει για τις ε, ε, τραπεζικές συναλλαγές, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ε, θέματα κεφαλαίων κλπ. Αυτά όλα είναι τμήματα των κοινών μας στόχων για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και βάσιμοι. Αυτό που έχουμε εδώ είναι το θέμα των ε, εποπτικών ελέγχων των ισολογικών πολιτικών για τους τραπεζίτες. Ε, με το χαμηλότερο των συλλαγών θυμάστε ότι τον Ιούλιο 2009 υιοθέτησε μια σχετική πρόταση Κομισιόν και πρόκειται για ένα τμήμα συνεχού προγράμματο για να εφαρμοστεί η εργασία της επιτροπή Βασιλείας για την επιτηρήση των τραπεζών. Η πρόταση αυτή τώρα τροποποιήθηκε στο Συμβούλιο. Θα το διαβάσετε φαντάζομαι το κείμενο του Συμβουλίου και ο στόχος είναι να αντικατοπτριστεί πάλι η εργασία της Επιτροπής Βασιλείας από τον Ιούλιο και σύμφωνα με τις ε, αρχές ε, τους ε, ομάδα εργασία επιτήρησης για τα χρηματοοικονομικά και βέβαια και με τις εργασίες της μας στο ε, πολλοί θεωρούν ότι δεν έχουμε τίποτα να πούμε στον τομέα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε κύριος η ενδυνάμωση των ε, κεφλικών απαιτήσεων για τα βιβλία τους, επανετυλοποίηση και η εισαγωγή συγκεκριμένων κανόνων και συμ... πραγματική ε, εποπτεία όσον αφορά τις μισθολογικές πολιτικές και επίσης τις ειδικές αποζημιώσεις. Τα μπόνια αυτά που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό και δημόσιο θέμα οπωσδήποτε είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπουμε ότι τύπος σήμερα λέει, ότι η, το κράτος ανέλαβε μια τράπεζα σκοταπώνους πουλ Ξέρετε ότι όλα αυτά είναι θέματα που θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας και να αντικατοπίσουμε στην έκθεσή μας. Η οδηγία έχει σαν στόχο να έχουν οι τράπεζες υψηλότερο ποσοστό κεφαλαίων και να αντικατοπτρίζει η εποπτεία μακροπρόθεσμη απόδοση, όχι βραχυπρόθεσμη. Μεγαλύτερες κεφαλογικές ε, απαιτήσει σημαίνει να προσέχουν καλύτερα τι επενδύσει κάνουν και σύμφωνα με την Επιτροπή Βασιλεία ε, χρειάζεται 11,5% συμπληρωματικό ποσοστό κεφαλαίου. Και όπως ξέρετε οι τράπεζες Ήρθαν πολλές εδώ σε μένα. Εγώ λέω όταν ήμουν ε, φοιτήτρια δεν μπορούσα να, να δω τον μάνατζερ στην τράπεζά μου για να μου δώσει ένα δάνειο. Τώρα έχω 20 έξω από το γραφείο μου περιμένουν ουρά. Και λένε ότι εάν αυξηθεί αυτό το ποσοστό του κεφαλικού αποθέματος θα έχει επιπτώσεις στην δανειοδοτική τους δυνατότητα θα χρειαστεί ένα 3 έως 4% συμπληρωματικό κεφάλαιο. Δεν είναι τόσο τραγικό λοιπόν όσο ε, αφήνουν να πιστεύουν ορισμένε οργανώσει του τραπεζικού τομέα. Επίσης, ανησυχούν ε, ε, οι τράπεζες για την ταχύτητα εφαρμογή στην ημερομηνία, δηλαδή 2010, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ γλίγορα και αυτό θα έχει επιπτώσει στην πραγματική οικονομία. Ε, ορισμένοι λοιπόν από τους λόγους αυτούς ζήτησαν μια σταδιακή εισαγωγή. Ε, μετά που θα υπάρξει παραδείγματο χάρη για τρία τρίμηνα αύξηση του ΑΕΠ. Η Κομισιόν θέλει να ε, εφαρμόσει τους κανόνες της Βασιλείας γιατί δεν έχουμε πολύ δυνατότητα εμείς να επιδράσουμε στην εικόνα που παρουσιάζεται όσον αφορά τις αρχές που έχουν ήδη συμφωνηθεί στη Βασιλεία και που είναι διεθνής, διεθνούς μορφής αλλά θεωρώ ότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κατά νου καλύτερους διακαιρισμούς και αν με υποστηρίξετε θα προσπαθήσω να δω που μπορούμε να ενδυναμώσουμε την εποπτεία του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό. Να μην δεχθούμε απλώς τις προτάσεις να τις εφαρμόσουμε χωρίς πραγματική εποπτεία από το Κοινοβούλιο. Για να δούμε τα θέματα που είναι πιο χωρίς, ε, χωρίς προβλήματα περισσότερο. Η πανεπιστημιοποίηση, παραδείγματος χάρη, και το CRD2 που σημαίνει νέοι κανόνες από τη Βασιλεία. Και υπάρχει μόνο μία σημαντική ουσιαστική διαφορά, δηλαδή η πρόταση Κομισιόν για προ, εκ των προτέρων έγκριση πολυπλόκων μεθόδων και πράξεων εφανατιτλοποίησης. Έτσι προβλέπεται από την Κομισιόν. και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα επιβληθούν σημαντικές κυρώσεις κεφαλουχικής μορφής. Στο, συμβούλιο του, στο κείμενο συγγνώμη του Συμβουλίου τα κράτη-μέρη διαφώνησαν πάνω γι' αυτό. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε κατά πόσον συμφωνούμε με την άποψη του Συμβουλίου ή κατά πόσον θέλουμε να επαναφέρουμε την άποψη της Κομισιόν. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Πάλι η ομάδα Βασιλείας επέβαλε κάποιες ε, διατάξεις το Σεπτέμβριο ε, φτάσανε μάλιστα σε συμπληρωματική ε, συμφωνία να αποκλείσουν κάποιες μορφές ε, συναλλαγών. αποφασίστηκε ότι οι μορφές αυτές που αφορούν άμεσα την πραγματική οικονομία και βιομηχανία δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Το λεγόμενο correlation trading θα πρέπει να εξαιρεθεί. Υπάρχει και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πάλι συμφωνούμε με την άποψη του Συμβουλίου ή έχουμε διαφορετικές απόψεις στον τομέα. Η Βασιλεία είπαν ότι θα πρέπει να εξαιρείται, αλλά υπάρχουν κάποιες ανησυχίε να επιτραπεί να αφήσουμε ελεύθερα στις τράπεζες στον τομέα Τη Οι είπαμε διακονοστές θα προτιμούσαν ένα ελάχιστο ε, κατόφλι κεφαλαίου. Ε, αυτό δεν θα συμφωνηθεί όμως, Βασιλεία, πριν ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, μελέτη μέχρι τον Ιούλιο. Γι' αυτό προτείνει το ε, Συμβούλιο ένα το όριο 8% και η Βασιλεία φαντάζομαι θα επιλέξει ένα όριο της τάξης του 5 με 10%. Ε, μου είπαν οι ε, ενδιαφερόμενοι ότι δεν συμφωνούν με το ο κατόφλι του 8% και λένε ότι ίσως θα ήταν τελικά περιττό γιατί η Βασιλεία ίσως τον Ιούλιο θα καταλήξει σε πιο χαμηλό όριο 5% φερειπίν. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί κύκλοι έχουν πρόβλημα με την ημερομηνία θέση ισχύ. Λένε ότι δεν μπορεί να γίνει μέχρι τα τέλη του 2010. Γιατί λένε δικαίως καμιά φορά ότι θα χρησιστούν ε, κάποιες εκατοντάδες ε, δισεκατομμυρίων ευρώ τους επόμενους μήνες και αυτό θα έχει επιπτώσεις στην δανειοδότηση. Και επίσης εξέφρασαν ανησυχίες ότι είπα δεν θα εφαρμόσει τις αλλαγές βασιλείας μέχρι την ημερομηνία εκείνη και θα υπάρξει τότε ένα πρόβλημα ε, μεταξύ των διαφόρων οικονομικών ε, χώρων. Αυτή δεν είναι η άποψή μου, είναι η άποψη που σας παρουσιάζω για να τη συζητήσουμε. Υπάρχουν ίσως και άλλα θέματα ε, που θα θέλετε να θέξετε. Άφησα το μισθολογικό θέμα τελευταίο. Εγώ πιστεύω ως πολιτικός ότι αναμένεται ως νομοθέτες να πάρουμε κάποιες έντονες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό Έχει γίνει πολλή δουλειά στον με αυτό. το Συμβούλιο για την Χρηματοπιστική Σταθερότητα δημοσίευσε το Σεπτέμβριο του 2009. Ε, δόθη το αποτέλεσμα αυτό στην ομάδα των G20 στο Pittsburgh και θα πρέπει να δούμε τώρα τι θα μπορεί να γίνει γιατί αυτό Τέσσερις οι έχουν επίπτωση στους μισθούς όλων εκείνων των οποίων οι αποφάσει μπορεί να έχουν επίδραση στις, ε, στο επίπεδο κινδύνου των άλλων ε, τραπεζών. Η αρχική κυβέρνηση, αντισταθμίσματα, ε, η δομή η μεσολογική, η παρουσία των στοιχείων και η εποπτεία. Τι έκανε η Κομισιόν η Κομισιόν εργάζεται πριν να υπάρξουν οι σχετικές προτάσεις και βασίστηκε στην έκθεση Λαροζιέρ που έλεγε ότι οι επασμίες αυτές να αντικατοπτρίζουν την απόδοση, να μην είναι εγγυημένες. Αυτή ήταν η βάση του μισθολογικού κειμένου στο πρόταση CRD 3. Υπάρχουν εκεί χρηματοπιστωτικά και μη χρηματοπιστωτικά ε, μέτρα. Η Κομισιόν καθορίζει μια σειρά ε, μέτρων. Θα πρέπει αυτό να προσαρμοστεί σύμφωνα με την EBA, με τη νέα ε, τραπεζική αρχή της Ένωσης και το Συμβούλιο προτείνει κάτι που πάει πολύ πιο μακριά. Έχει συγκεκριμένε λεπτομέρειε για τα μέτρα που αφορούν τι μισθολογικέ πολιτικέ, που αφορούν πάντα τι αποζημιώσει που δεν θα πρέπει να είναι εγγυημένε, αλλά να αντικατοπτρίζουν απόδοση. Το 50% θα πρέπει να μην πληρώνεται σε ρευστό, αλλά σε μετοχέ που θα πρέπει να κρατούνται οι μετοχές αυτές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 40% θα πρέπει να καταμερίζονται σε τρία χρόνια και οι συνάδελφοι πρέπει να αποφασίσουν τρία χρόνια είναι σωστό περιθώριο. Α, ορισμένο μου είπαν ότι όλες αυτές οι επενδύσεις είναι μακροπρόθεσμες, 5 με 7 χρόνια. Γιατί καμιά φορά είναι πολύ ψηλά τα ποσά αυτών των αποζημιώσεων και θα υπάρχει δυνατότητα μείωσή του, εάν η απόδοση του ατόμου ή τη επιχείρηση είναι πιο χαμηλή από εκείνη που προβλέπεται. Το Συμβούλιο είπε επίση ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις, ε, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα, το hedging για να αντικατο... αντιμετωπιστούν αυτές οι ε, αποζημιώσεις και αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει σε τακτά χρονικά διαστήματα ανακοίνωση προς το κοινό και η δημοσίευση των λεπτομερών πληροφοριών όσον αφορά τα χρήματα που δίνονται στους υψηλά ειστάμενους ε, των τραπεζών. Και θα πρέπει βέβαια να μην ε, αποδυναμώνει τη δυνατότητα ενός τραπεζικού οργανισμού υποζημιώσεις αυτές, να αυξήσει τη δυνατή δυνατότητα. Αυτά προς το παρόν. Μελετήστε το με την ησυχία σας. Κοίταξα όμως λίγο ε, τα κείμενα της ε, Κομισιόν, του Συμβουλίου και της Εποπτικής ε, Επιτροπής. Καμιά φορά το Συμβούλιο πήγε πιο μακριά, άλλες φορές δεν έχει προβλέψει τίποτα. Έκανα λοιπόν κάποιες επιλογές στο μέσο ο οποίος θεωρώ ότι το κείμενο του Συμβουλίου είναι πιο αδύναμο. Και τέλο, συνάδελφοι, μπορείτε ίσω να θέλετε να εξετάσετε τι γίνεται σε κάποια γιατί σε κάποια υπάρχει η δράση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει η εργασία πάρα πολύ. Στη Γαλλία επίση κάτι έγινε. Κάτω χώρε, Ελβετία, όλες έδρασαν ήδη. Στη Γαλλία, παραδείγματος το 5% της αποζημίωσης θα πρέπει να αναβληθεί στην πληρωμή του για τρία χρόνια και στη Γαλλία αυτό το ποσοστό που είναι σε μετοχές θα πρέπει να κρατηθεί δύο χρόνια τουλάχιστον. Ε, στην Ολλανδία δεν μπορούν να πάρουν αποζημίωση οι μάντατζερ αυτοί πάνω από το 100% του ετησίου τους μισθού. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες διαφορές. Το γεγονό ότι ορισμένα κρατημέλη έχουν ήδη κάτι αποφασίσει δεν σημαίνει ότι εμεί θα πρέπει να περιοριστούμε στα κείμενα που έχουμε μπροστά μας και για να τελειώσω έχω να σας πω ότι κάποιες από τις δημοσιοποιήσεις που έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι το 87% του κοινού θεωρούν ότι θα πρέπει να διακανονίσουμε ιδίω τι αποζημιώσει και τους μισθούς που πληρώνονται. Αυτό σημαίνει ότι είναι έντονη η ησυχία του κοινού και θα πρέπει κάτι να κάνουμε στον τομέα. Λοιπόν, σα έδωσα μια γενική εισαγωγή Οπωσδήποτε πολλά θα ξέχασα, πολλά θα θέλετε εσείς να παρουσιάσετε και θα σημειώσω ευχαρίστως τις ανησυχίες σας ή άμεσα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα ήθελα εγώ να προετοιμάσω γραπτή την πρόταση την επόμενη εβδομάδα για να τη στείλω στη μετάφραση να μπορέσει να ε, συζητηθεί στις 18 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, συνάδελφοι. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή απόψεων για τους ε, λόγους που αναφέρθηκαν ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την έκθεση έγκαιρα. Έχω λοιπόν στον κατάλογο των ε, μιλητών τον εαυτό μου που είμαι σκιώδη συγγήτρια για την Αλντε, την Πασκαλ Κάνταν και τον κύριο Μπούμαν που επίσης ζήτησε το λόγο. Και εκεί πρέπει να κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Εκτός ε, αν έρθει ο κύριος Κάρας αν έρθει ο κύριος ε, Κάρας, αλλιώς ε, ε, θα έλεγα να σας πάρουμε ως εκπρόσωπο του ΕΛΚ. Καθυστερήσαμε για 10 λεπτά γιατί δεν υπήρχε εδώ εκπρόσωπος του ΕΛΚ και γι' αυτό με μας πω ότι αυτή τη στιγμή, για να είμαι σας έχω βάλει λίγο στο μάτι. Δεν είναι προσωπικό τώρα αυτό, εντάξει το είπα για το ΕΛΚ. Φαντάζομαι ότι είχαν λόγο που απουσίασαν και δεν ήρθαν έγκαιρα. Όσον αφορά το CRD3, αυτό είναι ένα από τα πολλά μέτρα που θα ληφθούν και κατ' ουσίαν ε, αφορά τα αίτια της κρίσης. Δεν πρόκειται απλά για το ότι ε, θέλουμε να προστατεύσουμε τα κεφάλαια από μελλοντικού κινδύνους. Το γεγονός ότι τα χαρτοφυλάκια δεν είχαν καλυφθεί από επάρκεια κεφαλαίων, αυτό οδήγησε στο να ε, αναλυφθούν κίνδυνοι. Υπάρχει κάτι λοιπόν που δεν έχει τελειώσει και αυτό είναι πριν από την κρίση. Γιατί είναι γνωστό ότι οι κίνδυνοι των χαρτοφυλακίων ήταν γνωστή όπως ήταν και γνωστό το ότι υπήρχε πολύ μεγάλη έκθεση στο CRD2. Τώρα, η πρόταση που έχουμε μπροστά μας δεν αφορά και δεν καλύπτει όλο, όλα τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών. Πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι είναι δύσκολο να αλλάξουμε αυτή την πρόταση, αλλά οι συνάδελφοι έχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις να καταθέσουν. Επίσης πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια διαφοροποίηση κατά πόσον πρόκειται ε, για ε, ανταλλαγές ε, ακίνητης ή κινητής περιουσίας. Αυτό μπορεί στο μέλλον να ληφθεί υπόψη στα περίφημα τραπεζικά διαβατήρια. Ξέρω ότι πολλοί έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες για την αύξηση τραπεζικών κεφαλαίων τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη να δοθούν κονδύλια στην πραγματική οικονομία. Πάντως εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα αρχικής σημασίας γιατί έχει άμεση σχέση με τη συμπεριφορά και το ε, trading book, ε, το χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να ρυθμιστεί. Το CRD2 ε, ίσως αρχίσει να εφαρμόσει στο τέλος του 10. Πάντως ε, ήδη έχουμε χάσει κάποιο χρόνο το 80% αφορά τη συνθήκη της Βασιλείας 1 και θα τεθεί και αυτό σε ισχύ σε κάποιες χώρες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν κεφαλαϊκές ε, μετακινήσεις. Πριν τελικά λάβουμε μια απόφαση κατά πόσο η είναι σωστή ή όχι, θα πρέπει να έχουμε κατά νου μια σφαιρική εικόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, αμοιβέ, εγώ συμφωνώ σε γενικές γραμμές με αυτά που προτείνονται. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αυστηρότητα. Εγώ ε, δεν είμαι υπέρ των ΚΑΠΣ, ε, αλλά θεωρώ ότι είναι σωστό να έχουμε μια πολιτική απάντηση στα θέματα των αποζημιώσεων και όχι μόνο την εποπτεία. Το 22.8 του παραρτήματος 2 καταδεικνύει το σωστό τρόπο. Εκεί αναφέρεται ότι το κόστος του κεφαλαίου, ο κίνδυνος και η ρευστότητα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το να λάβει κανείς αυτά υπόψη αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί κόστος και να αντισταθμιστεί από κέρδος. Όμως εδώ δεν πρόκειται για κέρδος και δεν είναι σωστό να απευθύνεται σε κάποιον ε, που ε, δεν είναι εκείνος που έχει άμεση σχέση με το κεφάλαιο. Όταν ε, προκύπτουν κέρδη, αυτά επιμερίζονται διαφορετικά. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει κάποια αιτιολόγηση για, τις, για τα μπόνους, για αυτές τις πρόσθετες αμοιβέ, ακόμα και αν υπάρχει κάτι που αντιστοιχεί στο κόστος του ε, κεφαλαίου και στις πρόσθετες αμοιβέ αν δεν δοθούν αυτά τα χρήματα κάπου θα πρέπει αλλού να αναζητηθούν. Άρα δηλαδή υπάρχουν εδώ αποχρόντες λόγοι γιατί αν κάποιος ε, έχει παρουσιάσει μια καταπληκτική απόδοση αυτό ας πρέπει να ας ας γίνει γνωστό. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ε, γίνονται μεγάλα κέρδη και από ό,τι φαίνεται θα δοθούν και μεγάλα πριμ απλά και μόνο γιατί είχαμε χαμηλά επιτόκια ε, και ως εκ τούτου τα πριμ θα πρέπει να δίδονται για αποδόσεις που είναι πάνω από αυτό που προσφέρει η αγορά. Το να υπάρχουν περισσότερες αιτιολογήσεις, αυτό θα πρέπει να αφορά κυρίως ε, τα μεγάλα πριμ και όχι απαραίτητα τη μέθοδο με την οποία δίδονται αυτά τα πριμ. Εγώ δεν βλέπω γιατί να μην αναφέρουμε αυτούς ε, που τα λαμβάνουν. Γιατί να φοβόμαστε περισσότερο από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εγώ δεν πείθομαι από το επιχείρημα ότι αυτό ε, θα οδηγήσει στο να εγκαταλείψουν ε, οι άνθρωποι τις δουλειές τους ή ότι θα τους εκφοβήσουν. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ποιοι παίρνουν αυτά τα πριμ και ίσως ε, θα πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, όσον αφορά τη διάταξη για την τιτλοποίηση, ε, στο CRD2 γίνεται λόγος για την ε, τιτλοποίηση και η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι στο πνεύμα της αναλογικότητας που εισήγαγε το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την αμέλεια, την ολιγορία αυτή δεν προέρχεται από τη Βασιλεία 2, από αυτή τη συμφωνία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είτε θα θελήσουμε να συμφωνήσουμε με αυτά που έχουμε ήδη επιτύχει στη CRD2 ή να ακολουθήσουμε περισσότερο τη γραμμή του Συμβουλίου και να πούμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να εξετάζεται σε επίπεδο εποπτείας με τη νέα Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή η οποία θα πρέπει να θεσπίσει μια ολόκληρη σειρά κανόνων για το τι πρέπει να γίνει με πολλά θέματα. Υπάρχουν και άλλα, όχι μόνο η τιτλοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει μια καλύτερη δέσμη μέτρων που θα κατατεθεί. Εγώ ε, θεωρώ ότι όσον αφορά τις ε, συναλλαγές ε, γενικότερα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Εκείνο που πρέπει να αναγνωρίζουμε είναι ότι οι επόπτες θα πρέπει και αυτοί ε, να δίνουν το καλό παράδειγμα. Δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει απαραίτητα αυτή η δυνατότητα, ότι ισχύει αυτό απαραίτητα. Αυτές είναι οι δικές μου απόψεις προς το παρόν και ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου. Κοιτάξτε, ξεκινάμε με το θέμα των πριμ, των πόνους. Πράγματι, εδώ ε, γίνεται λόγος για πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν σε διεθνές επίπεδο έχει γίνει αρκετή δουλειά για, τις, για τα πρίμα αυτά τότε σε επίπεδο των G20 όσο και σε εθνικό επίπεδο και πολλά αντικατοπτρίζονται σε αυτά που λέει το Συμβούλιο. Κοιτάξτε, πολλοί ήρθαν και μου είπαν «Μα δεν πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη». Είναι ε, σημαντικά, εφόσον ε, υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και προσωπική ανέλυξη, η δυνατότητα αυτή. Σωστό αυτό, αλλά εγώ ε, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να δίδονται πριν που στο παρελθόν οδήγησαν ορισμένοι να αναλαμβάνουν πάρα πολλού κινδύνου ε, με τα χρήματα άλλων και τελικά αυτά ήταν τα χρήματα των φορολογουμένων. Εξάλλου αυτοί που υποτίθεται ότι κρατούσαν καλά στα χέρια τους εταιρείε, αυτοί που ήταν στα τμήματα χορήγησης πιστώσεων, αυτοί πολλές φορές αποζημιώνονται περισσότερο από τους κινδύνους που αναλάμβαναν και όχι από αυτούς που απέτρεπαν. Εντάξει υπάρχουν ε, μνήες αυτών των θεμάτων στις ε, αποφάσεις του ε, Συμβουλίου. Σε τελική ανάλυση δεν είναι οι θεσμοί που παίρνουν λάθος αποφάσεις, αλλά είναι τα άτομα που παίρνουν λάθος αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν και η αποζημίωση θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με άτομα. Διάφορα κράτη-μέλη εμφάνισαν τους δικούς τους τους κανόνες. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να μπορούν να εκπονούν τους δικούς τους τους κανόνες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια στάνταρτ πλατφόρμα για όλους. Παραδείγματος χάρη, το Βασίλειο είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να περιμένουμε του χρόνου, θέλουμε ε, να πούμε αυτό που λες και εσύ Σάρων, ότι ήδη εφέτος αρκετοί ε, θεσμοί ε, είχαν κερδοφορία και αυτό πολλές φορές με τα χρήματα των ε, φορολογουμένων. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη κατέβαλαν διαφορετικά ποσά. Μιλώντας όμως στον απλό άνθρωπο, εγώ πιστεύω ότι, και αυτό το πιστεύουν και οι φορολογούμενοι, ότι εκείνη είναι σε τελική ανάλυση οι ε, πιστωτές και γι' αυτό θα πρέπει οι ε, θεσμικοί επενδυτές και ο κλάδος γενικότερα να το έχουν αυτό κατά νου σε σχέση με τους κινδύνους. Αργότερα όταν θα μιλήσουμε για το φόρο των συναλλαγών, αν ο φορολογούμενος πρόκειται τελικά να συμμετέχει στις ε, ευθύνες τότε πολύ σωστά ο φορολογούμενος θα πρέπει και να ε, ζητείτε γνώμη του για τα χρήματα που δίδονται με τη μορφή πιστώσεων. Υπάρχουν εδώ κάποια πολύ σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με το σε ποιο σημείο αυξάνουμε την κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιον τρόπο προηγείται τη Συμφωνία Βασιλεία και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Εμεί χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για το χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών και επίση να είμαστε σίγουροι ότι μάθαμε το μάθημά μα από την τιτλοποίηση. Και στο μέλλον η τιτλοποίηση ε, δεν θα πρέπει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, αλλά να έχει μεγαλύτερη κεφαλαϊκή επάρκεια. Με τη γλώσσα της τιτλοποίησης υπάρχουν ανησυχίες ότι θα μπορούσαμε να εξαναγκάσουμε τις τράπεζες το αυριανό κεφάλαιο να το χρησιμοποιήσουν για τους κινδύνους των ε, λαθών του παρελθόντος. Έχοντας λοιπόν αυτά τα ε, επισφαλή, τοξικά δάνεια, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το μέλλον των τραπεζών και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κατάρρευση, αν θέλετε, στα κονδύλια για την πραγματική οικονομία. Μιλάμε δηλαδή για μέχρι και 150 δις, απλά και μόνο γιατί γίνεται λόγος για την τιτλοποίηση που αφορά στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι κάνει η Συμβολία της Βασιλείας για αυτή την αξιολόγηση. Τώρα, όσον αφορά το χαρτοφυλάκι και των συναλλαγών. Εδώ υπάρχουν τρεις διαφορετικές μορφές κεφαλαίου που προστίθενται. Ε, το παραδοσιακό μοντέλο ε, το κεφάλαιο κινδύνου υπάρχουν τρεις μορφές ε, κεφαλαίων που αυτές συνδυάζονται ε, μερικοί λένε ότι κάτω από ορισμένε συνθήκες αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένας, ε, ε, ένας θεσμικός επενδυτής θα μπορούσε να έχει περισσότερα κεφάλαια στο χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών από ό,τι στις τράπεζες. Αυτό θα ήταν λάθος να κρύβουν οι τράπεζες τα χρήματά τους και να μην παρουσιάζουν την πραγματική τους θέση. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε και αυτό κατά νου. Τώρα, η μελέτη αντικτύπων. Αυτό που αναφέραμε προηγουμένως για τα τρία κεφάλαια προστιθέντα, αυτό θα πρέπει να είναι μέχρι το 11,6 ε, του κεφαλαίου των τραπεζών στην Ευρωζώνη. Εγώ θέλω οι τράπεζες ε, να καλύπτουν το χαρτοφυλάκι των συναλλαγών με περισσότερα κεφάλαια, να αυξηθεί η κεφαλαϊκή επάρκεια. Μπορούμε βέβαια ε, να τι αναγκάσουμε να πάρουν το 2% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στην δανειοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν η Βασιλεία θα κάνει άλλη μία μελέτη αντικτύπων έχει ήδη ανατεθεί αυτή η μελέτη ε, τον Ιανουάριο υποτίθεται θα επανέλθουν και ανησυχώ γιατί πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να ακούσουμε τι θα μας πει η Συμφωνία της Βασιλείας και να διασφαλίσουμε ότι αν αυτοί τελικά αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν ότι θα πρέπει να ε, γίνονται οι δανειοδοτήσεις με βάση την κεφαλαϊκή επάρκεια, τότε καθοριστική είναι η συμφωνία της ε, Βασιλείας. Το ρυθμιστικό αρμπιτράζ ε, είναι και αυτό μεγάλη σημασία. Τελικά, αν αναγκάσουμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες να μειώσουν το μέγεθος των ισολογισμών τους, τότε αυτό θα είναι άλλο ένα χτύπημα, ένα κόλαφος για την Wall Street όπου οι ε, τράπεζες θα κληθούν πλέον να ε, καλύψουν τα κεφάλαια. Πρέπει να δούμε λιγάκι και την χρονική στιγμή της εμφάνισης αυτών των κεφαλαίων και να διασφαλίσουμε ότι δεν ε, διατρέχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλο κίνδυνο. Εγώ λέω να συνεργαστούμε με τη Συμφωνία της Βασιλείας, να δούμε τη μελέτη αντικτύπων και να είμαστε σίγουροι ότι όταν θα εισάγουμε τους κανόνες του αύριο, αυτοί δεν θα προκαλέσουν μία ρήξη ανάμεσα στα λάθη του χθες και την ε, δανειδιωτική πολιτική του αύριο, που θα έχει όμως άμεσες επιπτώσεις το σήμερα. Πασκάλ. Εσείς θέλετε το λόγο, είσαστε έτοιμος. Ας ακουστούν και λίγο γαλλικά στην αίθουσα αυτή. Δεν κάνει κακό η γλωσσική ποικιλομορφία. Πάντως δεν έχω να προσθέσω πολλά και πολύ συγκεκριμένα γιατί είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και δεν θέλω να μακρηγορήσω. Από πολιτικής απόψεως η ομάδα των Πρασίνων θα υποστηρίξει όλες τις προτάσεις από όπου και αν προέρχονται είτε από την Κομισιόν από το Συμβούλιο για να ενισχύσει να τον περισσότερο τον έλεγχο των ρίσκων που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Πιστεύω ότι σε αυτή την οδηγία μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία εις ό,τι αφορά τον έλεγχο των ιδίων πόρων και του λεγόμενου μοχλού αλλά βεβαίως και των ε, επενδυτικών ε, ταμείων που συνδέονται με το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα εφόσον είναι το πιο ε, επικίνδυνο με το μεγαλύτερο ρίσκο τέλο πάντων οικονομικό φαινόμενο. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε για την συλλογική χρήση της τιτλοποίησης των προϊόντων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ένας από τους λόγους της κρίσης, ότι αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούσαν παντού, κανείς δεν ήξερε τίποτα για αυτά. Ε, είχαν σήμανση 3α χωρίς να ξέρουμε τι κρυβόταν από πίσω και νομίζω ότι είναι απόλυτα θεμητό να απαγορευθεί, να απαγορευθεί η πολύπλοκη τίτλοποίηση και η επανατίτλοποίηση. Ε, άρα από αυτή την άποψη είναι εντελώς ανεπαρκής η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παρόλο που γνωρίζουμε ότι έχουμε περιορισμένε δυνατότητε Θέλουμε το κοινοβούλιο, ε, το κοινοβούλιο, αυτή είναι η επιθυμία μας, να μπορέσει να τροφοδοτήσει τη συζήτηση που θα οδηγήσει σε μία μελέτη των ε, πρακτικών δυνατοτήτων που έχουμε μετά από αυτή την κρίση. Ε, επιμένουμε πολύ για τα αρνητικά στοιχεία, αλλά δεν ασχολείται κανείς με τα θετικά. Ναι, γιατί υπάρχουν και θετικά μετά την κρίση με την έννοια ότι έχουμε μια ευκαιρία να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Τελευταίο σχόλιο. Σοκαρίστηκα, κυρία Μακάρθη, όταν σας άκουσα που είπατε ότι δεν ασπάζομαι τα λεγόμενα του τραπεζικού λόμπι, αλλά αναφέρω αυτό που μου είπαν οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα. Μα μόνο με τράπεζες μιλήσατε. Αυτό φαίνεται με αυτούς που εκπροσωπούν τις τράπεζες. Διότι εναλλακτικά δεν αναφέρεται τίποτα άλλο. Βεβαίως και να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι τράπεζε, αλλά εμείς ως νομοθέτες έχουμε υποχρέωση να ακούσουμε το σύνολο των κοινωνικών ε, δυνάμεων, το σύνολο των κοινωνικών παραγωγικών και οικονομικών ε, ε, δυνάμεων, αν μη τι άλλο για λόγους Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, λόγω του ότι έχει περάσει η ώρα και λόγω του γεγονότος ότι έπεται ευθύ αμέσω σε μία κρόση, θα εστιάσω την προσοχή μου σε δύο θέματα. Πρώτη παρατήρηση. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για, την, ε, για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το θέμα, με διαφάνεια και ακρίβεια. Νομίζω λοιπόν ότι η συγγήτρια είναι σε θέση να ορίσει ε, τα πρότυπα για το τι θα κάνουμε στο μέλλον με τις τράπεζες. Θα υπάρξει και άλλη έκθεση και εγώ θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να παραμείνετε σε αυτόν τον τρόπο που αντιμετωπίζετε πράγματα με αυτοπεποίθηση. Εμείς ε, δεν είμαστε ο βραχίωνας ε, των τραπεζών ούτε του Συμβουλίου ούτε της Συμφωνίας Βασιλείας. Εμείς είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα νομοθετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε με βάση αυτά που πιστεύουμε ότι είναι δίκαια και με τον τρόπο που πιστεύουμε ότι θα παρεμποδίσουμε την επόμενη κρίση. Την τελευταία δεν μπορέσαμε να την εμποδίσουμε γιατί δεν είχαμε νομική βάση. Και τώρα έρχομαι στη δεύτερη παρατηρήσή μου. Με πολύ μεγάλη έκπληξη άκουσα και θα πω μόνο αυτό, ότι όταν πρόκειται για ε, τις ε, τιτλοποιήσεις και τις ανατιτλοποιήσεις πρόκειται για πολύ περίεργα και περίπλοκα προϊόντα και ξέρουμε τι ρόλο έπαιξαν αυτά τα περίπλοκα προϊόντα στην κρίση. Έχουμε ακόμα στο νου μας ε, το τι έγινε, τα δράματα που προέκυψαν στις ε, τίτλοποιήσεις πλήρης ε, έλλειψη κατανόησης και δεν κατανοώ εγώ γιατί το Συμβούλιο λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια προέγκριση επανατιτλοποιήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω κυρία Πρόεδρε και εσάς, ε, κυρία Συγήτρια, την επόμενη φορά όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν, κυρίως για τα σημεία εκείνα όπου η πρόταση του Συμβουλίου αποτελεί ξεκάθαρα νόθευση της πρότασης Κομισιόν. Ε, κατά τα άλλα θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Κομισιόν. Ίσως σήμερα να μην έχουμε χρόνο. Νομίζω όμως ότι την επόμενη φορά μπορούμε να προγραμματίσουμε το να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν. Ε, κύριε Τιούρι, θέλετε να πείτε κάτι πολύ σύντομα. Ευχαριστώ και ελπίζω να μην το μετανιώσετε μετά την παρέμβασή μου που μου ζητήσατε να μιλήσω. Πρώτον, ε, γιατί θα είμαι σύντομη και δεύτερον, γιατί θα ήθελα να συμφωνήσω με κάτι που είπατε. Κοιτάξτε, το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω... Λοιπόν, ε, πρώτη ερώτηση. Με ακούτε? Υπάρχει διερμηνία. Μάλιστα, υπάρχει διερμηνία. Δεύτερη τώρα ερώτηση. Έχω να κάνω μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Γνωρίζετε κατά πόσον υπάρχει μελέτη αντικτύπων. Έχει διεξαχθεί τέτοια μελέτη που να έχει ερευνήσει τις ε, επιπτώσεις αυτών των μέτρων στην προσφορά πιστώσεων. Γιατί η κυρία Πρόεδρος ε, είπε ότι κατά κάποιο τρόπο έχει ρυθμιστεί το θέμα της ε, κεφαλαϊκής επάρκειας των τραπεζών. Αλλά ερωτώ, υπάρχει μελέτη αντικτύπου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί θα πρέπει το όλο θέμα να το δούμε και κάτω από το πρίσμα της ουδετερότητας του ανταγωνισμού. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία διοχετεύθηκαν ε, στους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αυτό δημιουργεί στρεβλό στην αγορά. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ήταν ε, παντού οι ίδιες οι ανάγκες. Έτσι λοιπόν, αν φτάσουμε στο CRD3 και στο CRD4 και ε, καταστήσουμε αυστηρότερους τους κανονισμούς για την ε, κεφαλογική επάρκεια, πρέπει να δούμε λιγάκι και το θέμα τι γίνεται με, την, με τον ανταγωνισμό. Γιατί ορισμένοι οργανισμοί έλαβαν πάρα πολλά χρήματα, αλλά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται, οι τράπεζες ήταν υγιέστερες, δεν είχαν μολυνθεί με τόσα πολλά τοξικά προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ερωτώ. Είναι δίκαιο να υπάρχει αυτή η φοβερή πρικοδότηση των ε, τραπεζών στην Δυτική Ευρώπη σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τα πριμ, θα περιμένουμε βέβαια το τέλος του έτους, αλλά πρέπει να σας πω ότι με πολύ μεγάλη ε, προσδοκία και ανυπομονησία περιμένω εδώ τι θα γίνει με τις πρόσθετες αυτές αμοιβέ, τα πριμ. Και θα μου επιτρέψετε και άλλη μια ερώτηση. Φαίνεται δεν έχουμε και πολύ χρονικό διάστημα στη διάθεσή μα. Ε, μιλήσατε για θέση ισχύ την άνοιξη 2010, μα δεν είναι και πολύ χρόνο. Φαίνεται ότι πρέπει να ε, προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που μου έδωσαν προσανατολισμού, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να εξετάσω ορισμένα από αυτά τα θέματα και να δω αν μπορώ να τα συμπεριλάβω. Θα ήθελα να καθισχάσω του πρασίνου ότι ε, δεν έχω συναντήσει και τόσο πολλού ενδιαφερομένου ε, αυτούς που έχουν προβλήματα ανέφερα, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη ότι αυτοί που έχουν προβλήματα είναι οι εκπρόσωποι του τραπεζικού κλάδου. Αυτό ήθελα να παρουσιάσω. Γιατί αυτοί έχουν πρόβλημα με τις προτάσεις αυτές. Είναι πολλοί άλλοι που δεν έχουν. Κυρία Φόρτ και θα τελειώσω με αυτό. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειε του ή άλλου κάποια στιγμή αργότερα. Είναι νομίζω ζωτική σημασία ζήτημα για την Επιτροπή αυτή και το Κοινοβούλιο. Θέλουμε να παρακολουθούμε απαθώς τις εξελίξεις στην παγκόσμια σκηνή ή θέλουμε να τις επηρεάζουμε. Θέλουμε να περιμένουμε το 2010 μέχρι να γίνει η αξιολόγηση της διαδικασία της Βασιλείας και μεταξύ να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Όχι. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Εμείς, εμείς θα πρέπει να ηγηθούμε της προσπαθίας αυτής και οι λοιποί να μας ακολουθούν και στο Οικονομικό Συμβούλιο και στις συναντήσεις μας με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία και με τις επισκέψεις μας στην Ουάσιγκτον να πείσουμε τους Αμερικανούς και άλλους ότι πρέπει αυτοί να ακολουθήσουν εμάς και όχι το αντίστροφο. Διότι αν υπάρξει και άλλη κρίση, ε, ποιος θα τα πληρώσει τα σπασμένα πάλι, ο φορολογούμενος, πάλι ο πολίτης και τότε θα έχουμε πρόβλημα. Αυτά πρέπει να προλάβουμε, αυτά πρέπει να προλάβουμε με τα κεφάλαια κινδύνου, με τα υπερβολικά μπόνους και τις αποζημιώσεις, και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που έθεσε η Πρόεδρος, των οποίων θα επανέλθουμε σε, αργότερο στάδιο, σε μεταγενέστερο στάδιο της συζήτησης. Αυτά ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη, διότι είχαμε πολύ λίγο χρόνο να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Η επόμενη φορά θα εξετάσουμε ε, το σχέδιο έκθεσης στις 26 Ιανουαρίου. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Ας ετοιμαστούμε τώρα για την ακρόαση. Και ζητώ συγγνώμη από το πάνελ των ομιλητών μας για την καθυστέρηση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομιλητές μας και να τους ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. προτείνω να ακούσουμε όλους τους ομιλητές, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνει ο καθένας την παρουσίασή του και μετά, και μετά να κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων και ένα γύρο απαντήσεων. Έχετε λάβει τα βιογραφικά των καλεσμένων μας δεν χρειάζεται να σας τους ε, παρουσιάσω. Οι ομιλητές μας θα πρέπει να περιοριστούν σε πέντε, άντε έξι λεπτά. Μεταδίδεται μέσω webstream η συνάντησή μας αυτή. και μετά τα αυτά να δώσω το λόγο στους ομιλητές με τη σειρά που έχω εγώ εδώ στο δικό μου χαρτί που ελπίζω να είναι η ίδια με αυτή που έχετε κι εσείς. Ο πρώτος ομιλητής είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ονομάζεται Αλεξάνδερ. Αλεξάνδερ, πώς το προφέρετε το επώνυμό σας. Βίντεο. Βίντεο. Παρακαλώ από τη Γενική Διεύθυνση Φορολόγησης και Τελωνιακής Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν εργαζόμαστε επί καμία συγκεκριμένης προτάσεως για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συζητάμε ατύπως και μεταξύ μας και με άλλους φορείς και θα σας αναφερθώ για την κατάσταση των πραγμάτων και για το που βρίσκονται οι συζητήσεις όχι μόνο στη δική μας ε, Γενική Διεύθυνση αλλά και σε άλλες ε, μονάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι θυμόμαστε τις συζητήσεις ε, για τον φοροτόμπιν, όπως τον ονομάζαμε παλιότερα. Τώρα είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μιλάμε για όλες τις ε, ή σχεδόν όλες τις ε, συναλλαγές. Για το πώς θα σχεδιαστεί ένας τέτοιος φόρος θα πρέπει να έχουμε κατά νου τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε. Το βασικό για μας είναι η συλλογή εισοδήματος για την παγίωση των δημοσίων οικονομικών των κρατών μελών. Το δεύτερο είναι να δούμε κατά πόσο ένας τέτοιος φόρος θα συνεισέφερε στην εξυγένση των παγκοσμίων οικονομικών και το τρίτο είναι να δούμε σε ποιο βαθμό η ο τραπεζικός κλάδος πρέπει να πληρώσει για τα λάθη του. Για την καλύτερη διαχείριση, για την καλύτερη διακυβέρνηση better regulation όπως λέμε σύμφωνα με τη δική μας ανάλυση με τα εφιστάμενα στοιχεία υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για τα αποτελέσματα ενός τέτοιου φόρου στις χρηματαγορές δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει την μείωση των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει την ε, σταθερότητα, την ρευστότητα, την διακύμανση των τιμών και ούτω καθεξής. Κάτι το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε μας οδηγεί θα έλεγα στο σαφές συμπέρασμα ότι δεν είναι το σωστό μέσο αυτός ο φόρος εάν θέλουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μας οδηγήσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για να το πω διαφορετικά. Εμείς είμαστε υπέρ μιας κανονιστικής προσέγγισης. Αυτή είναι η προτιμότερη. Μίλησα για το εισόδημα πριν και την φορολογική σταθερότητα και απαγίωση. Και τίθεται αμέσως το ερώτημα πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Στον εθνικό προπολογισμό, στον εθνικό κορβανά κατά κύριο λόγο. Αλλά συζητώνται και εναλλακτικέ λύσεις. Ανάπτυξη, περιβάλλον, ο κοινοτικό προπολογισμό, ο κοινοτικό κορβανάς. Δεν θα μπω πάντως σε λεπτομέρειες επ' αυτού. Θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι εξ όσων γνωρίζουμε η Ένωση και η Γερμανία θα συνεισφέρουν τα μάλα στην προσπάθεια αυτή, γιατί αυτές οι δύο αγορές είναι οι μεγαλύτερες. Και βεβαίως τίθενται θέμα δίκαιης κατανομής του βάρους, ε, επιμερισμού του εισοδήματο αυτού κτλ. Το V4, ένα αυστριακό Ινστιτούτο, έκανε κάποιου υπολογισμούς. 287 δι παγκοσμίω με συντελεστή 0,1% για την Ένωση 130 δις είναι το ποσό και συμπεριλαμβάνουμε εδώ όταν λέω Ένωση, Νορβηγία και Ελβετία. Ε, όχ, τέλος πάντων. Λάθος εδώ έχει διαφάνεια, δεν είναι τα δεδομένα το 2007 αλλά το 2006. Και θα έλεγα ότι είναι υπεραισιόδοξα τα στοιχεία αυτά. υπάρχει πτωτική εκτίμηση. Εις ό,τι αφορά την άμβλυνση των παρενεργειών, μείωση των εμπορικών ροών κτλ. Πάλι είναι υπερσιόδοξη η εικόνα που δίδεται μέσω αυτών των στοιχείων. τα οποία υπολογίζονται γενικώ με την συμπερίληψη όλων των αγορών. Είναι ένας μέσος όρος ας πούμε. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό διότι κάθε αγορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και οι διαφορές αυτές ε, το συνολικό, το η συνολική εικόνα δεν κατανέμεται ισόποσα ανά περίπτωση. Τι σημαίνει αυτό για το πώς θα πρέπει να οργανωθεί ένας τέτοιος φόρος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλήξουμε στην λεγόμενη κρίσιμη μάζα προϊόντων και γεωγραφικού εύρους. Μόνο η Βίφορ αυτό το Αυστριακό Ινστιτούτο έβαλε νούμερα και συμπεριέλαβε τις μετοχές και τα, τις χρηματιστριακές συναλλαγές, όπως επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία των χρηματοπιστωτικών φορέων. Φορολογική βάση τώρα. Αξία της συναλλαγής. Αλλά για τα παράλογα μιλάμε για ονομαστική αξία. Δηλαδή και το λανθάνον περιουσιακό στοιχείο της αξίας και όχι μόνο η αξία. Ο τομέας των παραγόγων λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει το μεγαλύτερη συνεισφορά εισοδήματο. Ο κίνδυνος μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η μεταγκατάσταση. Οι χρηματαγορές υπάρχει ο κίνδυνος να μετα, μεταγκατασταθούν σε άλλες περιοχές. Επίσης μπορεί να πληγούν οι επενδυτικές δυνατότητες των επιχειρήσεών μας και το δυναμικό τους για ανάπτυξη. Επίσης υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς προς προϊόντα που δεν υπόκεινται σε φόρο. Για τη γεωγραφική κάλυψη πρέπει να είναι ως δυνατόν ευρύτερη θα ήταν επικίνδυνο να καλυφθεί μόνο η Ένωση. Στο G20 συζητήθηκε, αλλά εκφράστηκαν πολλοί δισταγμοί, όπου σημαίνει ότι δεν είναι ρεαλιστική αυτή η προοπτική. Το Αυστριακό Ινστιτούτο προτείνει ως κριτήριο την ε, προτείνει ως κριτήριο την ώρα. Δηλαδή για την ώρα που κλείνει το χρηματιστήριο, οι περιοχές του κόσμου που έχουν την ίδια ώρα να συμμετέχουν σε αυτό το ε, σύστημα. Ας πούμε Greenwich, ώρα Greenwich. Τώρα, από νομοθετική απόψεως, δεν ξέρουμε μέχρι ποιο βαθμό είναι συμβατή αυτή η πρόταση με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Αλλά ε, υπάρχουν και άλλες νομοθεσίες που θα πρέπει να τροποποιηθούν για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Αυτά, εν συντομία, αυτά τα οποία ήθελα να σας αναφέρω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι απολύτω άδικο αυτό που κάνουμε, να σα περιορίζουμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Σα παρακαλώ όμω να το ε, προσπαθήσετε. Ο κύριος Τζεφ Λόιντ τώρα. Παρακαλώ εντός εξαλέπτου. Μια που δεν έχω PowerPoint εγώ, θα σας πω με δύο λόγια τι θέλω να σας πω. Μερικά εισαγωγικά σχόλια και ε, μετά κάποια σχόλια για τον ε, φόρο των ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Έχω να σας πω ότι ο ΣΑ δεν έχει εργαστεί πάρα πολύ πάνω στο θέμα των χρηματοοικονομικών φόρων. Και εγώ θέλω να σας τονίσω ότι μιλάω προσωπικά σήμερα, όχι εξ της ε, του Το θέμα βέβαια είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε, να υπάρχουν κάποια μέτρα για να καλύψουμε τα φορολογικά ελλείμματα που έχουμε προτείνω ότι φορολογικό αυτό παράγοντα θα μπορεί να είναι στη τάξη του 3% του ΑΕΠ. Δεν υπάρχουν βέβαια εύκολε λύσει και δεν υπάρχουν μεμονωμένε λύσει. Και οπωσδήποτε έχει από το ΩΣΑ. Εάν μια χρηματοπιστωτική κρίση έχει κάτι το θετικό και συνήθω οι καταστάσει έχουν κάτι θετικό, είναι η ευκαιρία που μα δίνει για να δούμε πού θα μπορέσουμε να ε, απλουστεύσουμε τους στόχους, να είμαστε πιο δίκαιοι και να αυξήσουμε και τα έσοδα. Γιατί συνήθως το πρόβλημα είναι ότι κοστίζουν μέτρα που υιοθετούνται, αλλά εδώ στο φορολογικό θέμα έχουμε οικονομικά ωφέλη. Σα έχει κάνει πολλά για την προώθηση της αλληλεγγύης της πληροφοριών διεθνώς και το έχει πετύχει αυτό με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν πολλές νέες συμφωνίες ανταλλαγής ε, πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η υπογραφή των συμφωνιών αυτών θα βοηθήσει οπωσδήποτε. Ίσως θα μπορούσε επίσης να εκταστεί το θέμα της αποφυγής ε, στο διεθνές τομέα για να πετύχουμε την αύξηση των εισοδομάτων. Περνώ στο κύριο θέμα που θέλετε να συζητηθείτε, οι νέε πηγέ χρηματοδότηση δηλαδή. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε νέα πηγή χρηματοδότηση θα πρέπει να ακολουθεί κάποιε βασικέ αρχέ. Θα πρέπει να είναι εύκολη και αποτελεσματική στη συλλογή τη, να μην κοστίζει πολύ, να είναι δύσκολο να αποφευχθεί. Θα πρέπει να είναι ουδέτερο όσον αφορά τι επιπτώσει στην οικονομία και τι ανακατάταξη, εκτός αν αυτός ήταν ο στόχος και τέλος θα πρέπει να ε, εξασφαλίσει την ε, αποδοχή των πολιτών. Ε, είναι σαφές ότι υπάρχει μια τροποποιημένη αντιμετώπιση της φορολογίας, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε την μεγάλη σημασία του χρηματοπιστωτικού τομέα για την πρόθεση της ανάπτυξης της οικονομικής. Υπάρχει λοιπόν κάποια μετα αντιμετώπιση της συζήτησης που αναφέρει τώρα κυρίως στο δυνατότητα του φόρου αυτού να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα. Υπάρχουν ακόμα δύο βασικά θέματα κατά τη γνώμη μου που θα πρέπει να εξεταστούν. Πώς θα ήταν καλύτερο να εστιαστούν οι φόροι αυτοί σε κερδοσοπικές ε, συναλλαγές και όχι πραγματικές χρηματοπιστωτικές ε, ε, συναλλαγές και θα πρέπει να γίνει αυτό και σε σχέση με την ε, αποδοχή από τους πολίτες και τη δυνατότητα αύξησης των εισόδων. Η Κομισιόν θεωρεί ότι το, το μεγαλύτερο τμήμα του φόρου αυτού θα προέρχεται από τα παράγωγα. Είναι δύσκολο να δούμε πώς θα μπορεί να εφαρμόσει το φόρο μάλλον σε κερδοσκοπικές και όχι τόσο σε μη κερδοσκοπικές ε, δραστηριότητες. Ε, συνήθως λέγεται βέβαια βραχυπρόθεσμο θα πει κερδοσκοπικό. Και ίσως αν επιβληθεί εκεί θα έχουν σημαντικότερες επιπτώσεις στις βραχυπρόθεσμες αυτές ε, συναλλαγές. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε και την δομή των αγορών. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες τύπου hedging και επίσης βραχυπρόθεσμες. Είναι βασικό το θέμα που σας είπα να δούμε πώς θα εστιαστούν οι προσπάθειες, ούτως ώστε τα... Ε, ο φόρος αυτός να εστιαστεί στα παράγωγα. Επίσης υπάρχει και το θέμα του ποιος τελικά θα φορολογείται, ποιος θα πληρώσει αυτό το φόρο. Παραδείγματος χάρη, όταν γίνεται μια μεταβίβαση ε, ε, ομολόγων ναι, γίνεται μεταξύ ατόμων που δεν κατοικούν σε μια χώρα, δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι ή δεν έχουν τη φορολογική του έδρα. Είναι λοιπόν δύσκολο να δούμε τι θα γίνει με το φόρο αυτό. Αυτά είναι κάποια θέματα σχετικά με τα παράγωγα. Υπάρχει ένα θέμα νομίζω που αφορά την ευρεία βάση του φόρου. Δηλαδή να εξασφαλιστεί τα προϊόντα να, μην μπορούν να καθιστούν από κάποια άλλο, η γεωγραφική τοποθέτηση να μην μπορεί να εργαστεί από κάποια άλλη. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι δραστηριότητε τι οποίε αναλαμβάνει η αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλέ βραχυπρόθεσμε ε, συναλλαγέ που γίνονται για την συνεχή προσαρμογή των χαρτοφυλακίων. Και ίσω τελικά η μορφή που υιοθετηθεί είναι διαφορετική, δηλαδή η χαρτοφυλάκια να μην ε, αλλά προσαρμόζονται τόσο γλίγορα και σημαντικά τα σε θα είναι εδώ οι επιπτώσει στα έσοδα. Πολλά λοιπόν θα πρέπει ακόμη να γίνουν για να εξαστεί τι θα πρέπει να γίνει. Σε γενικές γραμμές λοιπόν θεωρώ ότι αυτός ο φάκελος αξίζει να μελετηθεί. Υπάρχουν κάποια τεράστια θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όσα εξέτασε τον φόρο Τόρμπιν στο παρελθόν και ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικό πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των πηγών εισοδημάτων και κατά πόσον θα αναμειχθούν εδώ είναι θέμα των μελών μας, των μελών του ΣΑ. Θα δούμε κατά πόσον εμείς είμαστε εδώ στο σώμα για να εργαστούμε στην κατεύθυνση αυτή, οπωσδήποτε είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε. Και χαίρομαι να ακούσω συζήτηση σήμερα το απόγευμα εδώ. Πρώτα ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο Ξαβιερουλέ επικεφαλής υπεύθυνος για τη χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο γιατί ε, οι προηγούμενοι έφαγαν λιγάκι χρόνο. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου αναγνωρίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω αυτά που θα πω σήμερα να βοηθήσουν στις αποφάσεις που θα λάβετε. Βεβαίως έχουμε το δικό μας τον φόρο στην αλλαγών στο Ηνωμένο ε, Βασίλειο που αποκαλείται STEM Duty. Και ε, για να αναφερθώ λιγάκι και σε αυτά που είπαν οι ε, προλαλήσαντες που τα στηρίζουν επιφύλακτα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα των επιπτώσεων που είχε ο φόρος συναλλαγών ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στις ε, εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαϊκής επάρκειας. Αυτή τη στιγμή ε, έχουμε τον φόρο αυτό που επιβάλλεται σε 0,5% στις ε, κινητές αξίες ε, και σε κάποιες μετοχές. Εξάλλου πρόκειται για ένα φόρο που επιβάλλεται στην πραγματική οικονομία, φόρο που τον καταβάλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο οι ιδιώτες αποταμιευτές όσο και οι εταιρείε. Βεβαίως ο φόρος αυτός σε τελική ανάλυση ε, ε, δεν, πληρών, δεν καταβάλει το φόρος από τους ενδιάμεσους, είτε από τις εταιρείε είτε από τον τελικό καταναλωτή. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στις, ε, στα συμπεράσματα μιας μελέτης που υπολογίζει ότι ο φόρος αυτός μειώνει τις συναλλαγές κατά 20%. Αυτό απλά και μόνο που υπάρχει σημαίνει ότι αυξάνονται οι τιμές των μετοχών κατά 6,25%. Όλες ε, οι μετοχές, ε, μάλλον η ρευστότητα είναι καθοριστική σημασίας και ανάλογα με το ε, ποιος αποφασίζει, από εκεί εξαρτούνται και πάρα πολλά για την εξέλιξη των μεταχών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μία μελέτη που έχει καταρτιστεί μετά από γραπτή επερώτηση. Ο φόρος των συναλλαγών μπορεί να αυξήσει και την ε, πτυτικότητα. Στην πραγματική οικονομία έχουμε τις ε, εταιρείε και τους ε, καταθέτες που αναζητούν επενδύσεις. Το κόστος του κεφαλαίου για εταιρείε που αναζητούν επενδύσεις έχει αυξηθεί πάρα πολύ από το φόρο των συναλλαγών. Ο φόρος των συναλλαγών υπολογίστηκε ότι αυξάνει το, φόρο, το κόστος του κεφαλαίου κατά 4 μέχρι 12% ανάλογα με τον τομέα. Και οι μεγαλύτερες επιπτώσεις δυστυχώς υπάρχουν σε εταιρείε υψηλής τεχνολογίας. Το κόστο για του αποταμιευτέ και του επενδυτέ είναι σημαντικό. Στον Ηνωμένο Βασίλειο, φόρο συναλλαγών καταναλώνει το 3,5% τη αξία ε, των αποταμιεύσεων ε, ενός ε, μέσου πολίτη για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μειώνει το επενδυτικό κεφάλαιο στην οικονομία. Υπολογίζουμε ότι η κατάρριξη του στον Ηνωμένο θα οδηγούσε σε περίπου 6,4 δισεκατομμύρια λίρες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες επενδύσεις. Η έννοια του φόρου συναλλαγών αυτό ε, σημαίνει ότι αλλάζει κάπως ε, και η συμπεριφορά και γι' αυτό καταργήθηκε ο περίφημος ε, φόρος που αποκαλείται το τόμπινγκ. Η προϋπόθεση για αυτόν τον φόρο είναι ότι θα είναι αποτελεσματικός στο να καταπολεμά τις υπερβολές και κυρίως την υπερβολική δραστηριότητα στην αγορά. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπερβολική ρευστότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ ο τζίρος είναι περίπου το ένα δέκατο αυτού των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό προκύπτει κυρίως από εταιρείε μικρής και μεσαίας ε, κεφαλαϊκή επάρκεια. Οι μεγάλες μπορούν πάντα να βρουν επιπτώσει. Οι μικρές όμως δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Αν δούμε λοιπόν την αγορά των ΗΠΑ που έχει περίπου την ίδια κεφαλοποίηση όπως της Ευρωπαϊκής Ένωση, η ταχύτητα του κύκλου εργασιών είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Ευρώπη. Και αυτό προφανώ επηρεάζει την δυνατότητα των, κεφαλαίων, των εταιριών να καταφεύγουν σε κεφάλαιο και αυτό πάλι είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα για τις εταιρείε μικρής κεφαλαιοποίησης. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε στην Σουηδία όταν εισήχθη φόρος του 1% στις κινητές αξίες που διπλασιάστηκε αργότερα ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη και με την απόδοση των μετοχών και με τη ρευστότητα. Και γνωρίζουμε και από την Κίνα τον Μάιο του 2009 ε, τριπλασίασαν τον φόρο και μειώθηκε και ο τζίρος ε, στο χρηματιστήριο της Σανγκάης και η ρευστότητα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε ε, στο μέσο μιας μεγάλης οικονομικής ύφεσης η οποία προέρχεται από υπερβολική χρήση των πιστώσεων. Αυτό όμως μπορεί να προκύψει μόνο από υπερβολές που λαμβάνουν χώρα στις κινητές αξίες. Ενώ λοιπόν οι τράπεζες ε, ε, σήμερα καταφεύγουν στην αρνητική μόχλευση η ανάγκη να έχουν ε, διόρθωση των ισολογισμών τους τους οδηγεί στο να καταφύγουν σε νέα κεφάλαια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διατηρηθούν τα παραδοσιακά μέσα του να αποκτά κανεί κεφάλαιο από εκεί που υπάρχει είτε από ιδιωτικέ τράπεζες είτε από ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού οργανισμούς και αυτοί, ε, αυτά τα κεφάλαια να κατευθύνονται εκεί που χρειάζονται, κυρίως στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός ο φόρος των συναλλαγών κατ' ουσίαν τιμωρεί τη μόχλευση η οποία οδηγεί ε, κυρίως στις τράπεζες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό Σήμερα όπου όλοι αναζητούμε τρόπους για να προκαλέσουμε την οικονομική ανάκαμψη πρέπει να βρούμε δυνατότητες να διοχετεύονται περισσότερα κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η... Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαπιστώσει ότι οι επιπτώσει του φόρου συναλλαγών στην πραγματική οικονομία είναι ιδιαίτερα αρνητικέ. Πρέπει να αποφεύγουμε φόρου που μπορούν να ε, επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξάνεται το κόστος του κεφαλαίου για την πραγματική οικονομία και μακροπρόθεσμα ζημιώνεται η ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρος για να δεχθεί επενδύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σάνι Καπούρ, επόμενος ομιλητής, ε, ε, ο οποίος θα έχει ως θέμα τον αναπροσδιορισμό της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Δεν έχω παρουσίαση PowerPoint. Θα ήθελα να σας πω γιατί θα μιλήσω. Το πρώτο θέμα που θα αναφέρω είναι γιατί χρειαζόμαστε τον φόρο αυτό και εδώ είναι η σωστή πλατφόρμα για Και το δεύτερο είναι να διασκεδάσω κάποιες από τις ανησυχίες που έθεσαν διάφορες συνάδελφοι και το τρίτο τα πλεονεκτήματα αυτού του φόρου. Μετά τέταρτο θα μιλήσω για τις επικρίσεις και πέμπτο τι με λιγενέστε. Λοιπόν, ε, ζούμε παράδοξες, ε, παράδοξους καιρούς. Αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε οφείλεται κυρίως στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος έλαβε 3 δις δολάρια για να επιβιώσει από τον εθνικό, από το δημόσιο προπολογισμό. Τίποτα λοιπόν δεν άλλαξε, εκτός το ότι εμείς ε, οι κοινοί πολίτες έχουμε κάποια προβλήματα ε, απασχόλησης, ανεργίας ε, και απώλειας εισοδήματος. Έχουμε και ρεκόρ φορολογικών ελλημάτων. Δε και η σταθερότητα στην Ευρωζώνη απειλείται. Τι έγινε με την Ελλάδα, τι έγινε νωρίτερα με την Ιρλανδία. Πρέπει να βρούμε εισόδημα λοιπόν, φορολογικό. Από πού θα προέλθει. Δεν είναι κανονική η καιρή, όπου θα αρκούσε δηλαδή απλώς να αυξήσουμε το φόρο. Η ανάγκη για φορολογικό εισόδημα είναι απόλυτα σαφής. Από πού θα έρθει. Από την αύξηση του ΦΠΑ. Θα ήταν καταστροφικό γιατί θα αποθάρρυνε την κατανάλωση. Θα μπορούσε να έρθει από το φόρο εισοδήματο. Αλλά αυτό θα έπλητε την παραγωγή. Θα μπορούσε να προέλθει και από έναν τύπου τόμπιν φόρο. Ένας φόρος κανείς δεν θα πει ναι είναι καλή ιδέα, τον δεχόμαστε, παρακαλώ περάστε να μας τον επιβάλλετε. Το θέμα είναι ποιον θα φορολογήσουμε, τον καταναλωτή, τον εργαζόμενο ή τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτές είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Αυτή λοιπόν δεν είναι η καλύτερη, αλλά είναι η λιγότερο κακή. Το μη χείρον. Κάποιος μίλησε για ευκαιρίες που προέκυψαν από την κρίση. Κάτι το οποίο φάνηκε σαφώς είναι η πολυπροκότητα του όλου συστήματος του συστημικού κινδύνου, της οργάνωσης, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των σχετικών αγορών. Υπάρχει ένας τρόπος ε, να πλήξουμε, να μειώσουμε δηλαδή την ε, πολυπλοκότητα και άρα το συστημικό κίνδυνο. Επίσης, ο βραχυπρόθεσμος ορίζοντας, το εύκολο κέρδος είναι κάτι που θα πρέπει να παταχθεί. Όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση, όταν οι χρηματιστές, οι brokers είναι μηχανές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Όταν ε, τα, τα κομπιούτερ ε, απέτυχαν παταγωδός λόγω έλλειψης ανθρώπινης κρίσης να μετριάσουν τη φιλοδοξία του κέρδους είδαμε τα πρώτα σημάδια αυτής της κρίσης. Τεχνητά φούσκωσε, μεγάλωσαν οι όγκοι των συναλλαγών και μετατοπίστηκε το κέντρο, το κέντρο ε, βάρους από μια μακροπρόθεσμη προοπτική επένδυσης προς ένα βραχυπρόθεσμο κέντρο. Αυτοί οι υπολογιστές πολλές φορές ε, βρίσκονται ε, πολύ κοντά, φυσικά κοντά στους, στους μεγάλους, στα μεγάλα κέντρα αποφάσεων, ας πούμε στο City, είναι δίπλα στο χρηματοστήριο. Λίγα δευτερόλεπτα αρκούν Λίγα δευτερόλεπτα αρκούν για να γίνει στρέβλωση ανταγωνισμού. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, ε, το δυναμικό του εισοδήματος είναι τεράστιο και με εντυπωσίασαν πολύ ε, τα αριθμητικά στοιχεία που έδωσε ο κύριος ε, από το αγγλικό χρηματιστήριο. Δηλαδή, αν μιλάμε για 0,5% είναι πολύ, πολύ καλό, πολύ υψηλός φόρος. Τώρα, ε, δεν νομίζω ότι θα στεγνώσουν ε, οι αγορές, ότι δεν θα υπάρχει δηλαδή ρευστότητα. Άρα είναι πολύ καλή ιδέα αν είναι έτσι όντως τα πράγματα. Αν είναι 3 με 6% μακροπρόθεσμα, μην ξεχνάμε ότι από το 1600, 400 χρόνια ισχύει αυτός ο φόρος στο Ηνωμένο Βασίλειο και μακροπρόθεσμα ε, μείωσε 3 ε, με 6% τις πληθωριστικές τάσεις. Τη φούσκα δηλαδή. Ε, γιατί, γιατί να είναι κακό δηλαδή αυτό. Ίσα ίσα εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ καλό. Αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα προσμετράται στο σωστό, του, της πλαίσιο. Δηλαδή, τι μπορεί αυτός ο φόρος να προσφέρει ως εισόδημα σε σχέση με τις άλλες δυνατότητες που υπάρχουν. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάποια πλεονεκτήματα των φόρων αυτών. Είναι εύκολος, είναι ηλεκτρονικός, συλλέγεται εύκολα ε, οι νέοι κανονισμοί για την κεντρικοποίηση των παραγόγων, για τα clearing houses και για την ε, καταγραφή όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, για την ρύθμιση όλων των χρηματαγορών, όλων των δικαιοδοσιών. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο φόρος θα είναι αδύνατο να τον αποφύγει κανείς, είτε τον εφαρμόσει μονομερός, είτε παγκόσμια. Επίσης είναι ενδυνάμει και σταθεροποιητικός παράγοντας για τη συναγορά, το ανέφερα. Οι επικρίσεις ότι είναι δηλαδή δυσαναλογικός, ότι θα προβλήματα στα διευθυντικά ταμεία, ότι θα μειώσει τη ρευστότητα στις αγορές, ότι θα αυξήσει την πτυτικότητα, δεν ισχύουν. Είναι υπερβολικά πράγματα τα οποία βεβαίως είναι απολύτω αναμενόμενα από τον κλάδο. Um, Σας ευχαριστώ. Ο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανένας μετά από τέσσερις τόσο διακεκριμένους ε, εμπερευνόμενες. Θα κεράσω τρία κύρια θέματα. Ποιοι είναι οι στόχοι των φόρων αυτό, ποια είναι τα ενδυνάμει προβλήματα και ποιες είναι οι ενδεχόμενες αναλλακτικέ των φόρων από το χρηματικό κόστο στην Γιατί άμα δούμε το ποια είναι τα θετικά στοιχεία, θα πρέπει να σκεφτούμε και τα προβλήματα που υπάρχουν. On the one hand here you see possible objectives and of course the list. Ε, βέβαια ο πίνακας δεν είναι πλήρης, κάθε άλλο. Από την άλλη μεριά βλέπετε εδώ κάποια ενδεχόμενα μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Το πρώτο θέμα που θα μπορέσει κανείς να ρωτήσει κατά πόσον είναι σαν ένας ε, σουηδικός σουλιάς αυτός ο φόρος. Δηλαδή, ξέρετε, αυτός ο, ο, ο, ο ελβετικός ε, μπορεί να κάνει τα πάντα. Ή μήπως και αυτός ο φόρος το ίδιο είναι. Πρέπει να ρωτήσουμε. Είναι ε, μια χρήσιμη προσθήκη στα άλλα εργαλεία που υπάρχουν. Και θα κάνω κάποιο έτσι εν μέρει πολιτικό και εν μέρει τεχνικό σχόλιο. Αναλυτικά το θέμα, όπως δεν είναι κατά πόσον ο φόρος αυτός είναι καλύτερος από το να μην κάνουμε τίποτα. Είναι κατά πόσον είναι πραγματικά πιο κατάλληλος για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν από άλλα ενδεχόμενα ε, μέσα. Η κύρια σύγκριση είναι μεταξύ του φόρου από το χρηματοκρατών συναλλόγων και άλλων μεθόδων που μπορούσε κάποιο να επιλέξει. Για τους πολιτικούς εδώ είναι σαφές ότι δεν μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν όλα τα ενδεχόμενα μέσα μέσα στα πλαίσια του, σημερινού, του σημερινού συγγνώμη, πολιτικού πεδίου. Εάν παραδείγματο ήταν η τρίτη καλύτερη λύση αυτό ο φόρο για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά ήταν σαφέ ότι η καλύτερη και η δεύτερη καλύτερη λύση ήταν πολιτικά απαράδεκτη ή όχι διαθέσιμη, ενώ ο φόρος από των χρηματοπιστωτικών ήταν ευρέως διαθέσιμη, θα έπρεπε να επιλέξουμε αυτήν την τρίτη καλύτερη λύση. Ε, πανεπιστημιακή όμως ε, αλήθεια θα έλεγε ότι αυτή όμως δεν είναι καλύτερη λύση και η τελευταία λύση έχουν και οι δύο δίκαιο. Και αυτό που έχει καταστήσει τη συζήτηση δύσκολη και ενδεχομένω επικίνδυνη είναι ότι ορισμένοι ερευνητέ δεν δέχονται την πολιτική διάσταση και πολιτικοί πολλές φορές δεν δέχονται την ευθύνη των ε, αναλυτών και των εμπειρογνωμών που λένε ότι αυτή η λίστα ήταν καλύτερη αν γίνει πρακτικά εφαρμόσιμο. Και η μεν και η ιδέα δηλαδή κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, η σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών τρόπων σκέψης θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν τόσα διδάγματα από την κρίση από εκείνα που ήθελαν είτε οι εμπειρογνώμες ή οι πολιτικοί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Θα αναφερθώ τώρα λίγο περισσότερο στην... δεν θα τα εξετάσω όλες αυτές τις, ε, αυτά τα, τα, σχέδια. Θα περάσουμε τώρα σε διάφορα παραδείγματα εθνικών φόρων επί των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν είναι τώρα θα τελειώσουν ε, επειδή υπάρχει ένας τέτοιος φόρος. Ακούσαμε για το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι ένα μεγάλο κέντρο χρηματοπιστωτικό παρόλο που έχει ένα φόρο πάνω στις συναλλαγές. Γίνεται λοιπόν αυτό. Βέβαια η δυστυχής εμπειρία ήταν όπως ξέρετε από τη Σουηδία που εισήχθη ένας φόρος των συναλλαγών αυτών που δεν ήταν καλά προετοιμασμένος, δεν, δεν εισήχθη σωστά μειώνεται η ρευστότητα. Τώρα το 20% δεν ξέρω είναι πολύ, είναι λίγο, τι να σας πω, μειώνουν πάντα τη ρευστότητα. Και το θέμα είναι κατά πόσο είναι καλό ή όχι. Εκείνο που είναι αντίθετο προς τον φόρο αυτό των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, λένε ότι η μείωση αυτή τη ρευστότητα θα μειώσει την αποτελεσματικότητα των αγορών, θα, ε, θα αυξήσει συγγνώμη, την επιτυχότητα και θα πλήξει την οικονομία. Άλλοι όμως είπαν ότι δεν έχει πολύ καλή χρήση ε, η κοινωνία για κερδοσκοπικές ε, δραστηριότητες και το υψηλό τους επίπεδο θα μειωθεί. Και η πτυτικότητα ίσως δεν, εφαρμ... δεν παρουσιαστεί τόσο πολύ. Εμπειρικές όμως αυτές ε, δηλώσεις δεν είναι και τόσο αποτελεσματικές. Υπάρχει το θέμα της επίπτωσης στο κόστος χρηματοδότησης. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που ακούσαμε ότι ο φόρος αυτός θα οδηγήσει σε μια πτώση των ε, τιμών των μετοχών και έτσι θα χρειαστεί περισσότερο κεφάλαιο, άρα θα είναι πιο ακριβό το σύστημα. Ταυτόχρονα όμως θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος της διαχείρισης του κινδύνου για μη χρηματοπιστωτικές εταιρείε θα ήταν πιο δύσκολο να ε, πωλήσει κανένας ε, τον κίνδυνο αυτό, το ρίσκο αυτό και έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη αποχή από ε, την ε, ανάληψη τόσο υψηλού κινδύνου. Αλλά η εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο είδε ότι δεν υπήρχαν σημαντικότατες επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας. Υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά. Θα πρέπει να δούμε όμως κατά πόσον περισσότερα είναι τα πλεονεκτήματα από ότι το κόστος. Υπάρχουν προβλήματα αποφυγής ε, και διαφυγής δεν θα σας το αναπτύξω αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα περάσουμε στην τελευταία διαφάνεια. Το πραγματικά σημαντικό σημείο είναι ότι η κρίση ήταν μια κρίση εμπιστοσύνης. Και γι' αυτό έχουμε μια μεταφορά όσον αφορά το βάρος απόδειξης. Γιατί πριν από την κρίση θα λέγαμε είμαστε επιπισμένοι ότι ο φόρος απάνω στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές είναι η καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε και η απάντηση θα ήταν όχι. Σήμερα όμως περισσότεροι λένε είμαστε επιπισμένοι ότι ο φόρος αυτός δεν θα πρέπει να είναι ένα τμήμα των εργαλείων που χρησιμοποιούμε μετά την κρίση. Δεν μπορούμε να πούμε ε, ναι, μπορεί πραγματικά να έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει ο φόλο αυτό πάνω στι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Παραμένει όμω αρκετή αβεβαιότητα, όπω ακούσαμε. Εδώ θέλω να κλείσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα χάρηκαν πάρα πολύ. Δεν έχει τελειώσει γιατί μου πατάνε εδώ το κουμπί να μιλάτε λίγο πιο αργά, να βοσβήνει το λαμπάκι. Δεν έγινε τίποτα. Έχω λοιπόν τέσσερις ε, βουλευτές που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας ε, θα τεθούν όλες οι ερωτήσεις και μετά ε, θα δοθούν οι απαντήσεις. Άλλος παρακαλώ. Κανείς άλλος. Η Κάθριν. Μία ερώτηση γενικής φύσεως είναι μία απάντηση σε γραπτή ερώτηση Κομισιόν τον Ιούλιο για το ενδεχόμενο της πανευρωπαϊκού φόρου χρηματικών συναλλαγών. Η Κομισιόν στην γραπτή της απάντηση λέει ότι ασχολείται με το θέμα αυτό ενός τέτοιου είδους πανευρωπαϊκού φόρου, όμως η Κομισιόν είναι επιφυλακτική ε, με την εισαγωγή αυτού του φόρου γιατί υπάρχουν και οικονομικές και νομικές επιφυλάξεις. Και ε, παρακάτω αναφέρεται ότι ε, δεν έχουμε καταλήξει υπάρχουν κίνδυνοι που εμπλέκονται με την εισαγωγή ενός τέτοιου φόρου. Ο φόρος ε, θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος κεφαλαίου για τις ε, εταιρείες. Γι' αυτό λοιπόν αν δεν υπάρξει μια παγκόσμια δράση τελικά θα είναι μια πράξη στην Ευρώπη με μισή καρδιά. Και ρωτώ τους ομιλητές, συμφωνείτε ότι το να λάβει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέτρο αυτό θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και στη τελική ανάλυση ε, ποιος ε, θα αποφασίζει πότε και πώς θα διανέμονται τα κεφάλαια. Ευχαριστώ πολύ. Τρει ερωτήσεις έχω να κάνω. Ε, μία παρατήρηση και δύο ερωτήσεις κατ' ουσίαν. Δηλαδή, αν μπορούμε να... Εφόσον διαπιστώνουμε ότι ο όγκο συναλλαγών είναι περίπου το 70 πλάσιο του παγκόσμιου ΑΕΠ και αν ποτίθεται γνωρίζουμε ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η αγορά η λανθασμένη αυτή η δόμηση της αγοράς είναι κατ' ουσίαν το αίτιο το γιατί η οικονομία μας διατρέχει τη χειρότερη κρίση από το 29-30. Αν ισχύουν λοιπόν όλα αυτά, τότε έχει νόημα να πούμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από, το, από τη βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία και να περάσουμε σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Πρέπει δηλαδή να προτιμήσουμε τον επενδυτή μακράς πνοής, ο οποίος κάνει επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο. Αν όλα αυτά λοιπόν ισχύουν, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ε, θα έπρεπε να γίνει μια, ένας νέος επιμερισμός ε, των ε, πόρων. Και αν γίνει τελικά να γίνει με μακροπρόθεσμη προοπτική. Τώρα απευθύνομαι στους εμπειρογνώμονες. Συμφωνείτε εσείς ότι πράγματι χρειαζόμαστε αυτή τη διάρκεια στις επενδύσεις. Αν πείτε ναι και δεν θέλετε όμως από την άλλη τα κείμενα, τότε πέστε μας ποια είναι η εναλλακτική λύση. Τι περιμένετε για να προωθήσετε το μακροπρόθεσμο στοιχείο. Αν πείτε ότι είστε κατά των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, τότε παρακαλώ πολύ να μας το αιτιολογήσετε. Και υπάρχει και ένα δεύτερο αντεπιχείρημα, το οποίο προβάλλεται επανειλημμένα, ότι αν τελικά εισαχθεί αυτός ο φόρος, θα προκύψει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι υπέρχημαχοι όμως λένε ότι αν αυτό τον φόρο τον βάλουμε στην ίδια ζώνη χρόνου, ε, δεν θα προκύψουν οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού, γιατί τι γίνεται, οι κερδοσκοπίες θα γίνονται την ίδια ώρα, την ίδια χρονική στιγμή. Και θα ήθελα να έχω κάποια απάντηση σε αυτό το θέμα, γιατί στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο βέλτιστο μέγεθος του φόρου και σε ποια ακριβώς γεωγραφική ζώνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις ε, παρεμβάσεις τους. Έχω ένα σύνολο ερωτημάτων να θέσω. Μιλάμε για ένα φόρο που μπορεί να εφαρμοστεί, ενό νέου φόρο που μπορεί να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχει κάποιος υπολογισμός των διοικητικών δαπανών που θα επισύρει αυτός ο φόρος. Διότι οι διοικητικέ αρχές σε κάθε κράτο μέλο έχουν ε, διαφορετικές συνήθειες ε, και παραδόσεις, ε, διαφορετικές υποχρεώσεις κτλ. Λοιπόν, έχει γίνει κάποια μελέτη, έχει γίνει κάποιος υπολογισμός για το κόστος το διοικητικό. Δεύτερο, ο φόρο αυτό συμμορφούται με μία από τι βασικέ αρχέ της φορολογίας που είναι η αρχή της απλότητος. Πρέπει να γίνεται απλά η συλλογή αυτού του φόρου. Είναι δυνατόν αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τρίτο, πώς συμμορφούνται, πώς ε, μπορεί αυτό να συνδυαστεί με την κατάσταση των offshores. Φόρος και ύπαρξη offshore σημαίνει ότι πρημοδοτούμε τις offshore που δεν δίνουν πληροφορίες και που έχουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων εκτός νομιμότητος ουσιαστικά. Τέταρτο, ισχύει ή όχι ότι ένας τέτοιος φόρος θα έχει ακριβώς την ίδια συνέπεια με το ίδιο αποτέλεσμα με τον ΦΠΑ. Όποιος πληρώνει το φόρο στο κράτος δεν είναι αυτός που πλήττεται από τις παρενέργειες ή την φοροδιαφυγή ή την φορολογική απάτη. Είναι αυτός που κερδίζει, ενώ αυτός που πλήττεται είναι ο τελικός καταναλωτής. Και τέλος, και με αυτό ολοκληρώνω, ένας τέτοιος φόρος δεν είναι ουσιαστικά μια κύρωση και αν ναι, γιατί να επιβάλλουμε την κύρωση και να τελειώνουμε, συγγνώμη για την έκφραση δεν θα είχε αυτό πιο σταθεροποιητικό χαρακτήρα, η κύρωση και αποτρεπτικό χαρακτήρα από την ένας φόρος. Πρόεδρος, επειδή πιέζει ο χρόνος θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις και θα απαντήσετε με μιας, γιατί αλλιώς δεν θα, περάσουμε, δεν θα προλάβουμε να περάσουμε σε δεύτερο γύρο. Χωρίς μικρόφωνο, παρακαλούμε. Λοιπόν, στη δική μου τη χώρα, τη Γερμανία, έχουμε μία εκπομπή στη τηλεόραση, το Pro Contra. Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Παρουσιάζεται μία υπόθεση και ακούγονται τα υπέρ και τα κατά. Οι Υπέρμαχοι και οι πολέμοι. Και σήμερα ήταν μια θαυμάσια συνεδρίαση αυτή που είχαμε, ε, γιατί ακούσαμε και τα υπέρ και τα κατά. Ο κύριος Φων Βάιτσέκερ ήταν ε, ε, από τη μία πλευρά και οι υπόλοιποι από την άλλη. Ε, βλέπω λοιπόν, καταλήγω στο εξή. αυτή η εμπειρική προσέγγιση δεν μας βοηθάει να προχωρήσουμε εμπειρικά δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο κατά πόσο η εισαγωγή αυτού του φόρου θα σημαίνει τον κατακλυσμό ή κατά πόσον θα σωθεί ο κόσμος. Κύριε Γόλε, εσείς ε, μιλήσατε ε, για το STEM Beauty, για αυτό το φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό όμως είναι άδικο γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος. Δεν μπορούμε να πάρουμε ως βάση το 0,5% και να συγκρίνουμε τις επιπτώσεις αυτού του 0,5% με τις επιπτώσεις ε, που θα έχει ένας φόρος του 0,01%. Άρα δηλαδή καθαρά εμπειρικά αυτό για μένα δεν είναι σαφές και σε τελική ανάλυση δεν θα μας απομείνει τίποτα άλλο παρά να κατανοήσουμε την εισαγωγή μη του φόρου ως πολιτική απόφαση. Και τι θα γίνει αυτό που έγινε πριν από κάποια χρόνια στη Γερμανία. Οι σοσιαλδημοκράτες ξεκίνησαν την προεκλογική εκστρατεία και είπαν μηδέν αύξηση φόρων. Οι χριστιανοδημοκράτες κατέβηκαν στην εκστρατεία και είπαν 2% αύξηση φόρων. Και όταν έφτιαξαν το μεγάλο συνασπισμό, τι κάνανε, αύξησαν το ΦΠΑ κατά 3%. Εμείς θέλουμε να τα αποφύγουμε αυτό. Και τίθεται λοιπόν το εξή ερώτημα. Αν τελικά είναι, πρόκειται για πολιτική απόφαση που θα ληφθεί μόνο αν είμαστε απόλυτα σίγουροι για το ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να επιτύχουμε με αυτό το φόρο και οι στόχοι ποιοι είναι. Θέλουμε να φέρουμε τάξη στα δημόσια οικονομικά ή μήπω στόχο είναι από το παραθυράκι να εισάγουμε τον πρώτο πανευρωπαϊκό φόρο, κάτι που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Θα το βάλουμε αυτό από την Κερκόπορτα ή μήπω θέλουμε να εφαρμόσουμε τον επιμερισμό του βάρους ή και πάλι μήπως ε, θέλουμε να συμπεριλάβουμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, σε αυτές τις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή. Αλλά αν δεν συμφωνούμε για τους στόχους, τότε είτε τον εισάγουμε, είτε δεν τον εισάγουμε το φόρο, περί το να συζητάμε. Η Κάθριν. Κάθριν Στάιλα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η εσπερίδα μας αυτή. Θα είμαι σύντομη. Ορίζουμε το φόρο αυτό με τον ίδιο τρόπο. Εννοούμε όλοι με τον αυτό τρόπο την έννοια αυτή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως ό,τι φορά τις εναλλακτικές. Θα με ενδιαφέρα ε, πολύ να ακούσω την άποψη των ομιλητών. Ποια είναι η εναλλακτική για την επίλυση ενός προβλήματος που είναι αντικειμενικό. Ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα. Αν υπάρχει τέτοιο φόρος και αν δηλαδή ο χρηματοπιστωτικό τομέα, οι χρηματαγορέ συνεισφέρουν με τον τρόπο αυτό στην κάλυψη κάποιου κομματιού των συναλλαγών. Το ποσό θα είναι τεράστιο. Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία μαζί είναι 97% του συνόλου των συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό για να αποφύγουμε και αυτό που είπε κάποιος ομιλητής ότι θα πρέπει αλλιώς να αυξήσουμε το φόρο εισοδήματος ή το συντελεστή ΦΠΑ που είναι και πολιτικό επιχείρημα. Ο κύριος Φαν Βαϊτσέκερ είπε κάτι για το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση ή σε αντιμολία με τη Σουηδία. Μπορείτε να μας το ξαναεξηγήσετε γιατί δεν το κατάλαβα πλήρως. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα η κυρία Μακάρθη. πολιτικά θα πρέπει να δεχθούμε ότι έχει οριμάσει η ιδέα αυτή, ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. 53% της κοινή γνώμης είναι υπέρ ενός κάποιου φόρου για τις συναλλαγές. Και 43% των συντηρητικών της κοινή γνώμης των συντηρητικών ψηφοφόρων. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο παραβίασε η χρηματαγορά. Παραβίασαν οι χρηματαγορές. Και υπάρχει ανησυχία για το ποιος θα πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απαντήσεις. Είναι ερωτήματα όμως ενδιαφέροντα. Και το G20, να μην ξεχνάμε, ότι ανέφερε και κάποιες άλλες ιδέες ας πούμε ένας φόρος επί των ασφαλιών, των ασφαλίστρων και ο φόρος για τις συναλλαγές ήταν μία από τις εναλλακτικέ. Αλλά η ομάδα των 20, το G20, ανέφερε πολλές άλλες εναλλακτικέ. Δεν ισχύει ότι μπορούμε να ανοιχνεύσουμε αυτούς τους φόρους σχετικά εύκολα επειδή έχουν κεντροποιημένο χαρακτήρα. Δεν ισχύει ότι ένας τέτοιος φόρος για τις συναλλαγές ουσιαστικά αν τον είχαμε επιβάλει από παλαιότερα θα είχε ως αποτέλεσμα την πρόληψη αυτής της κρίσεως. Και θα πρέπει να έχουμε κατά νου το στόχο. Και επιμένω το κοινό είναι σαφώς υπέρ αυτής της ε, λύσεως. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ακόμα ομιλητές. Γκίγκολτ, Χάνσπετερ Μάρτιν και Γκέτ Έτινγκ Παρακαλώ σύντομα, διότι αλλιώς θα ακούσουμε τις ερωτήσεις σας, αλλά όχι τις απαντήσεις του πάνελ. Καταρχήν, έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, άκουσα με ενδιαφέρον ότι ο ΣΑ και η Κομισιόν δεν αντιμετωπίζουν το θέμα με μια πρώτη στην εξέταση τι είναι δυνατόν να γίνει. Γιατί ε, μια από πολλές χώρες ε, συμπεριφέρθηκαν θετικά, δεν θέλω να ξέρω πότε θα προετοιμάσετε ή θα αρχίσετε τουλάχιστον να προετοιμάσετε νομοθετικά μέτρα, μια από τόσες χώρες μέλη αντιδρούν θετικά, θα πρέπει να προετοιμαστείτε και όχι να συλλέγετε αντιεπιχειρήματα. Μια πρώτη ερώτηση, ιδίως προς τον κύριο Βίντεο. Δεύτερον, Απορώ που στις παρουσιάσεις κυρίως ακούσαμε για ένα μοντέλο του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αλλά να δείτε μια απόφαση του ε, Κοινοβουλίου στην Αυστρία που αναφέρεται στο μηχανισμό ΣΠΑΝ και αυτός ο μηχανισμός είναι αντίθετος προς τις τάσεις των ε, της ανίδρασης αγέλης που υπάρχει. Και αυτός ο μηχανισμός θα ήταν ένα μέσο αντιμετώπισης του και γι' αυτό θέλω να ξέρω την άποψή σας. Και τέλος, αναρωτιέμαι το εξή. Εν ώψη του τεράστιου δυναμικού εσόδων, αναρωτιέμαι λέω ποιες είναι οι εναλλακτικέ και στη σκέψη σας κατά να εξετάζεται πόσο θα κοστίσει τα διεθνή αυτά χρηματοδοτικά αγαθά να μην διατίθεται ελεύθερα. Τέλος, μία παρατήρηση το γεγονός ότι οι φόροι αυτοί θα μεταβιβάζονται δεν σημαίνει ότι θα μεταβιβάζονται ε, αυτόματα σε όλους. Και αυτό το λέω με μεγάλο ενδιαφέρον του, προς τον κύριο Κλίντς που είχε την εντύπωση ότι για τις τοπικές αγορές σε μια χώρα ε, προτιμά τις τοπικές αγορές θα πληγεί από το φόρο διαφορετικά από μια χώρα που εργάζεται στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Και δεν άκουσα λοιπόν εγώ κάτι σχετικό στις συμβολές του πάνελ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χάσπιτε Μάρτιν. Ευχαριστώ, θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος. Και εγώ απόρρισα για τον τρόπο με τον οποίο ο επιχειμα... παρουσίασε τα επιχειρηματά του εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Ο κύριο Λόιντ είπε ότι ήταν προσωπικέ οι παρασυρήσει που έκανε. Γιατί νομίζω ότι μια που η κατάσταση στα κράτη με είναι τόσο ενδιαφέρον, θα έπρεπε κύριε Βίντο να πείτε ότι είναι πολύ προσωπικό αυτό που λέτε. Γιατί ε, παρουσιάσετε πιο πολιτικά τα θέματα από ότι πολλοί από τους βουλευτές. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι για ένα μεγάλο τμήμα των εμπειρογνωμόνων και αυτό να πάρει μια ερώτηση προς τον κύριο Βίντο αναφέρθηκε ότι υπάρχει δυνατότητα της επιβολής του φόρου αυτού σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο στο παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήθελα να μου το αναλύσετε αυτό κατά πόσον αυτοί που δεν εκφράστηκαν από αυτού θεωρούν ότι αυτή είναι μια δυνατότητα. Αλλά δεν μπορώ παρά να τονίσω αυτό που και ο Αν σα. Εάν αυτό δεν είναι ένα μέσο για να περιοριστούν κερδοσκοπικές στάσεις, τι αξίζει από την άποψή σα και τι θα ήταν μια καλή εναλλακτική για αυτό το στόχο. Ευχαριστώ κύριε Σέπεριν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όποτε ακούω το Αρμπίν, φόρος σκέφτομαι το τέρας του λοχνέ, γιατί θυμάμαι πριν από 6 χρόνια συζητιόταν το ένα ε, το ίδιο θέμα και τότε εγώ ήμουν στην Κομισιόν. Τώρα έχουμε το αδελφό του, του φόρου Τόρμ, που είναι το FTT, αυτό ο φόρο τη κροπιδοτικές Εγώ θα έλεγα ένα φόρο που δεν χρειαζόμαστε, δεν πρέπει να τον έχουμε. Γιατί θα πρέπει να έχουμε αυτό το νέο φόρο για φορολογική παγίωση, όπω είπαμε μπορεί κανένας να προσαρμοστεί και το εύρος του κράτους για να φτάσουμε εκεί. γι' αυτό το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε για αύξηση των εισοδημάτων, για την ε, στην εργασία των, στην ανάπτυξη. Δεν νομίζω γιατί ο κ. Στούφερ που είναι υπεύθυνο για την αναπτυξιακή συνεργασία λέει ότι ο προορισμό του δεν λειτουργεί σωστά. Δεν λειτουργεί λοιπόν το σύστημα. Για το περιβάλλον έχουμε πολλούς πράσινους φόρους για τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό, μα δεν θα έπρεπε να έχουμε έναν ε, προπολογισμό που θα μπει από την πίσω πόρτα. Ο κ. Λαμπάλατ είπε ότι θέλει να κόψει το, να περικόψει μάλλον το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 5%. Πολύ ενδιαφέρον μου φαίνεται. Λοιπόν, αυτό ο χώρο εδώ δεν μου φαίνεται ότι χρειάζεται. Αυτό το τέρας του Λοχνές ελπίζω να εξαφανιστεί το γλυκόρο των δυνατών. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Πολύ σαφή αυτά. Θα σα δώσω το λόγο αντίστροφα. Οι έσονται πρώτοι. Και σα παρακαλώ να απαντήσετε. Ο κύριο Φων θέλει να πάρει το λόγο πρώτος. Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε κάποιε ερωτήσει να τις ε, δώσετε στου συνάδελφου να απαντήσουν. Θεωρώ ότι ένα από τα ερωτήματα που επαναλήφθηκε συχνά. Είναι το θέμα της κρίσης του φόρου αυτού και πώς όλα αυτά συσχετίζονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω το ερώτημα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Φερρυπίν ιδέα να χρησιμοποιηθεί ένας φόρος για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές για να χρηματοδοθεί η αναπτυξιακή βοήθεια το ξέρετε σίγουρα. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα αποτυχιών και είναι πολιτικές αποτυχίες όταν ένας φόρος συσχετίζεται με μια δαπάνη που έχει επίσης αδύναμη πολιτική υποστήριξη. Αυτό νομίζω είναι η συνταγή αποτυχία. Εάν ήθελε κανένας να κάνει κάτι τέτοιο, ένα εθνικό δηλαδή φόρο χρηματοδοτικών συναλλαγών θα ήταν πιο ασφαλές αυτό το φόρο που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο που οδηγεί σε σημαντικά έσοδα για το κράτος. Αυτό είναι πιο ασφαλές. Γιατί ακριβώς τα έσοδα πάνε στον γενικό προπολογισμό του κράτους. Εάν πανούνται για κάτι άλλο, ενδεχομένως εκτός της χώρας, θα υπήρχε πολιτική πίεση σήμερα να εξαλειφθεί αυτός ο φόρος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα θέμα που αφορά την πολιτική οικονομία. Και η εξήγηση που έχω για την, το συζητισμό αυτό μεταξύ πολιτικά ευαίσθητου προγράμματος ε, για φόρους και πολιτικό ευαίσθητου ευάλωτων ε, στόχων και αυτό που αναφέρετε εσείς είναι, ναι, είναι ότι εκείνοι που είναι υπέρ θεωρούν ότι είναι θαυμάσια γιατί αυτά τα δύο συνενώνονται και μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου. Εκείνοι που είναι κατά όμω δεν εξάπτονται. Λένε άσους να μιλάνε, δεν έγινε τίποτα. Και αν κανένας ήταν πολύ σοβαρός γι' αυτό θα έπρεπε να αρχίζει να μελετάει τον συσχετισμό πολιτικά ισχυρό λόμπι για δαπάνες. Ε, κάτι τέτοιο έγινε στη Γερμανία. Πρόκειται για το φόρο στο πετρέλαιο. Η αύξηση του φόρου ε, για το πετρέλαιο ήταν πολιτικά ευάλωτος. Αλλά όταν συσχετήθηκε με το να αυξηθεί αυτός ο φόρος για να μην μειωθούν οι συντάξεις. Όλοι οι συνταξιούχοι ήταν υπέρ λοιπόν, οπότε ο φόρος πέρασε. Αυτό νομίζω σας παρουσιάζει και κάθαρα αυτό το σημείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το έχουμε κατά νου. Επίσης υπήρχε μια ειδική ερώτηση που μου υπευλήθη για το θέμα του Ηνωμένου Βασίλειου έναντι Σουηθίας. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασίλειου αυτό το λεγόμενο stamp duty σχετίζεται με τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας. Θα μπορούσε κανείς να φέρει τις μετοχές αυτές ε, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και να περάσει περισσότερο. Αλλά για ορισμένου ε, τύπους ε, τέτοιων πωλήσεων εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ο φόρος που εμβάλλεται είναι τριπλάσιος. Στη Σουηδία ήταν πολύ πιο εύκολη η αποφυγή του φόρου. Να πει, ας πούμε, θα κάνω τις συναλλαγές μου στο Λονδίνο. Έγινε αυτό. Και δεν υπήρχε αρκετός φόρος που συλλέγεται στην Σουηδία. Λοιπόν, ο τρόπο με τον πληρώνει το φόρο αυτό και πώ έχει οργανωθεί έχει σημαντικότητα τι επιπτώσει στο κατά πόσο είναι δυνατόν να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που είναι σαφέ και σχετίστηκε με κάποιε από τι άλλε ερωτήσει που υπευλήθησαν. Αυτό που είναι σαφέ λέω ότι όσο πιο πολλέ χώρε συμμετέχουν, τόσο πιο εύκολο είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τη αποφυγή και τη διαφυγή του φόρου. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στο παρελθόν ήταν δυνατόν να συλλεχθούν σημαντικά εισοδήματα στο εσωτερικό μιας χώρας. Δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε, γιατί όπως αναφέρθηκε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεγάλη αγορά και συλλάγει πολύ εισοδήματο. Ε, η Γερμανία σε ορισμένους τομείς έχει μεγάλες αγορές. Το υπόλοιπο όμως τη Ευρώπη δεν νομίζω ότι θα συλλεχθούν και τόσα πολλά χρήματα. Πρέπει να κάνεις πολύ προσεκτικό σχετικά για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι προβλήματα να μιλήσουν, θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σκαπόρ. Uh, thank you very much. Uh, let me also start by addressing... Λοιπόν, επιτρέψτε μου ε, να ξεκινήσω αναφερόμενος πρώτα απ' όλα στην ουσία του θέματος που είναι η ρευστότητα. Όσον αφορά την απόδοση της αγοράς, να είμαι σαφής, η απόδοση της αγοράς, μάλλον ο τζίρος δεν είναι το ίδιο όπως η ρευστότητα. Μπορεί κανείς να έχει μια αγορά με πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών και πολύ περιορισμένη ρευστότητα. Η ρευστότητα προέρχεται από τη διάσταση απόψεων. Όταν εγώ θέλω να πουλήσω, κάποιος άλλος θέλει να αγοράσει. Και πολύ συχνά αυτή αυτό το μοντέλο, το βραχυπρόθεσμο που βασίζεται σε τεχνικούς κανόνες, δηλαδή που λέει αγόρασε όταν πέφτουν τιμές και πούλησε όταν είναι ψηλά, αυτό επιτείνει τη ρευστότητα. Ε, η μείωση του κύκλου εργασιών του Λονδίνου δεν έχει σχέση με τη ρευστότητα. Είναι πολύ πιο περίπλοκο το μοντέλο, είναι διαφορετικό, είναι ένα μοντέλο το οποίο πολλές φορές είναι άμεσα συνεδεμένο με το σύνολο των συναλλαγών στην αγορά. Και αναφερθώ και σε κάτι άλλο που υπόθηκε, ότι πέντε φορές μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα που μετακινούνται οι μετοχές στις ΗΠΑ από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, έτσι είναι, γιατί εδώ υπάρχει ένα μοντέλο για επιχειρήσεις. Αυτό είναι το βασικό μοντέλο στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις περισσότερες κοινωνικές χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε για μια τελείως διαφορετική βάση και μοντέλο αγοράς. Δεν σημαίνει ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο σύστημα. Αυτό αυτό είναι το αποτέλεσμα επιλογών και δομών. Και να διευκρινίσω και ένα τρίτο στοιχείο. Αναφέρθηκε ότι όταν εισήχθη ο φόρο αυτό των συναλλογών στην Κίνα, μειώθηκαν οι μετοχέ, οι τιμέ των μετοχών κατά περίπου 20%. Κάτι τέτοιο. Μετά όμω από μια εβδομάδα, αν το δει κανεί, κάθε φορά που έπεφταν οι τιμέ ε, όταν εισήγεται αυτό ο φόρο, μετά αναπηδούσαν, ξανανεβαίνανε. Ακόμα και πιο ψηλά από το επίπεδο που ήταν. Άρα δηλαδή το επιχείρημά σα είναι έολο. Τώρα, όσον αφορά τη Σουηδία, ε, ο φόρος στη Σουηδία ήταν ε, πολύ κακά σχεδιασμένος, ήταν σαν να ε, ζητούσε να καταστρατηγηθεί και συνέβη μετά. Επίση που θέλω να πω ότι ακόμα και ένα κακά σχεδιασμένο ο αποδίδει έσοδα και η νέα ρυθμιστική ατζέντα που συζητείτε ε, θα καταστήσει την αποφυγή πολύ πιο δύσκολη. Ένα άλλο θέμα που ετέθη είναι το εξή. Ποιο θα πληρώσει τελική ανάλυση αυτό το φόρο, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική ερώτηση. Το γεγονό είναι ότι αν δει κανεί ε, το άκρο δεξιό του φάσματο, τον Φρίντμαν, κάποιον τέτοιο, αυτοί λένε δεν έχει νόημα να φορολογεί κανεί τι επιχειρήσει γιατί σε τελική ανάλυση η επιχείρηση μετακυλεί το κόστος του φόρου στους καταναλωτές, σωστό ενδεχομένω, ή ο φόρος πηγαίνει στους επενδυτές. Και αυτό είναι αλήθεια. Και όλοι αυτοί είναι άτομα. Κάθε μεμονωμένος φόρος στον κόσμο κάποια στιγμή είτε είναι φόρο πετρελαίου είτε εταιριών αεροπορικών ή ΦΠΑ εμείς τα πληρώνουμε αυτά το θέμα είναι ε, πώ πώς εξελίσσεται ο φόρος προοδευτικά ή ε, μειωτικά προς τα κάτω αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν δείτε ποιο επενδύει στα hedge funds ε, ε, ποιος επενδύει με υψηλή συχνότητα αυτό περνάει μέσα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και φτάνει μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο εδώ μέσα. Και πρέπει αυτό να είναι πολύ πιο προοδευτικό από το να αυξηθεί το ΦΠΑ ή ο εταιρικό φόρο ή ο φόρο εισοδήματο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου. Σε τελική ανάλυση, τα άτομα, οι πολίτε είναι που πληρώνουν το φόρο. Είναι καθαρά και μόνο θέμα ε, επιμερισμού. Υπάρχει το θέμα του ανταγωνισμού. Κατά πόσον, ε, εάν υπάρχει μόνο φόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό κατά πόσον θα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά τη. Κοιτάξτε, η ζώνη χρόνου δεν είναι σημαντική, γιατί αν θέλει κανεί να παραβιάσει κάτι, αυτοί στι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να κερδίσουν εκατομμύρια αν μείνουν ε, τη νύχτα ξύπνοι. Και αν μπορούν οι νυχτοφύλακε να κερδίσουν εκατομμύρια, γιατί να μην μπορούν οι επενδυτέ. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Σημασία έχει το νόμισμα. Εάν υπήρχαν επιθέσεις σε συναλλαγές στην Ευρωζώνη, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί όλα θα έπρεπε να γίνονται κάτω ε, ή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ίδιο και σε σχέση με άλλες αγορές. Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς ακριβώς ε, παγιώνονται οι λειτουργίες ε, της αγοράς, πώς ε, θωρακίζονται με νομοθετικές διατάξεις. Υπάρχει και το ερώτημα κατά πόσον ε, το κόστος του συντονισμού θα είναι υψηλό ή όχι. Αν το συγκρίνουμε με άλλους τόξους, παραδείγματος χάρη με εταιρικού ε, φόρους που οδηγούν σε μεγάλο βαθμό σε φοροδιαφυγή, αυτός είναι πολύ πιο απλό από όλους για να εφαρμοστεί. Γιατί όλες οι συναλλαγές είναι ηλεκτρονικές, καταγράφονται με στάνταρτ πρότυπο, ε, το, message, το μήνυμα δίνεται SWIFT και το κόστος συγκέντρωσης και το κόστος του συντονισμού είναι πολύ πιο χαμηλό από οποιαδήποτε άλλη μορφή φόρου η που υπάρχει. Η κίνδυνη για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αποφάσισε να τον εφαρμόσει τον φόρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν πρέπει να έχουμε το κόμπλεξ ότι είμαστε κατώτεροι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος κάποιος ε, να κινδυνεύει να μην έχει εδώ παρουσία γιατί για να μην έχει ένα φόρο 0,01% ή έστω παραπάνω. Είναι αδύνατον αυτό να συμβεί και με τους ε, νέους ε, κανονισμούς αλλά και με τους ισχύοντες είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος χώρος στον κόσμο που θα εφάρμοζε αυτό το φόρο. Ναι, πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμη προοπτική. Αν κάνει κανείς συνέντευξη σε μάνατζερ στη Νέα Υόρκη ή διευθύνοντα στελέχη ε, πολύ συχνά λένε και μπορείτε να το τσεκάρετε αυτό λένε λοιπόν ότι πολύ συχνά δεν κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις γιατί βραχυπρόθεσμα ε, θα τιμωρηθούν από τις αγορές που είναι βραχυπρόθεσμα προσανατολισμένες. Έτσι λοιπόν το μακροπρόθεσμο αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα και διότι έχουμε δει τα προβλήματα που ανέκυψαν με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν εσωτερικοποιούμε, παραδείγματο το κόστο τη κλιματική αλλαγή. Δεν απορροφούμε το κόστο των συντακτικών προβλημάτων. Άρα δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο φόρος αυτός είναι πολύ καλός. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία όπως ε, παραδείγματος χάρη είναι να εκπίπτει από ε, κεφαλαιακά κέρδη, αλλά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τελειώνω, τελειώνω σιγά σιγά. Πραγματικά ήμουν πολύ γενναιόδορη. Αν αφήστε λίγο χρόνο και για τους άλλους. Λοιπόν, τέλειωσα. Αυτά. Επόμενος. Φαντάζομαι ότι δεν θα συμφωνείτε με τίποτα από αυτά που ακούσατε. Και εγώ για τον ε, κοινοπολίτη θα ήθελα να μιλήσω. Μιλώντας για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο 280 χρόνια υπάρχει το χρηματοδοτηστήριο του Λονδίνου. Όχι 400 που είπε κάποιος, 280. Έχουμε και άλλο παράδειγμα. Με το Ιταλικό χρηματιστήριο. 4, κάτι δις συναλλάσσει σε blue chips. Αλλά με κεφαλοποίηση το... η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι τριπλάσια. Υπάρχει λοιπόν τεράστια διαφορά. Και αυτό είναι εις βάρος των επιχειρήσεων. Όταν ψάχνουν κεφάλαιο, αλλά δεν ζημιώνει την BP και την Glaxo και τα μεγαθύρια όσο επηρεάζει τις μικρές επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρχει ρευστότητα αρκετή για τις τεράστιες επιχειρήσεις, φανταστείτε πόσο δεν υπάρχει για τις μικρές, που είναι αυτές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, εάν θέλουν ρευστότητα θα τη βρουν εύκολα ή δύσκολο. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ακούω ότι το stamp duty είναι 0,5 ενώ ο φόρος το είναι 0,01. Η πρόεδρος, η κυρία Μπόλτς, είπε ότι δεν μιλάμε για το φόρο Tobin που είναι το 0,01 αλλά έναν φόρο για τις ε, χρηματοπιστωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο συντελεστής δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ποσοστό την έννοια συζητάμε την αρχή επιβολής ενός τέτοιου φόρου φυσικά και το stamp duty με 0,5% είναι εξαιρετικά υψηλό, αλλά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ποσοστό αυτού του νέου φόρου. Το θέμα είναι αν, ε, έχει, αν επιφέρει εισόδημα ή όχι. Αλλά ο, το, ο, ο φόρος δεν ε, έχει αυτή την ε, λειτουργία. Δεν έχει αυτό τον προσανατολισμό. Δεν πρόκειται για το εισόδημα. Και αυτά που λέει ο κύριος Καπόρ α, ε, ως α, ε, κοινός άνθρωπος, στο κάτω-κάτω όλοι κοινοί άνθρωποι είμαστε. Ο φόρος λοιπόν συνδέεται με την έννοια της κύρωσης. Θέλουμε να βελτιρίσει των χρηματαγορών ή θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε νέες μορφές φορολόγησης των επιχειρήσεων. Αλλά ας μην αυταπατώμεθα. Η κρίση προέρχεται από το επιθετικό στυλ με το οποίο συμπεριφέρεται ο τραπεζικός τομέας σε συνδυασμό με μια ρυθμιστική αποτυχία, δηλαδή την αποτυχία ελέγχου. Αν ο στόχος είναι να τιμωρήσει κανείς αυτό το τελευταίο, τις δομές της αγοράς που αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές, ε, δεν μπορεί να το ε, ε, επιτυχεί έτσι. Αφήστε που δεν θα σμειωθούν οι τράπεζε και οι διαμεσολαβητέ, θα σμειωθούν οι, τράπεζε, οι μικρέ επιχειρήσει, συγγνώμη, που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν, να βρουν του απαραίτητου πόρου. Α μην συγχαίουμε το μοχλό, τι τράπεζε, τι χρηματαγορέ και τη δομή των χρηματαγορών. Είναι διαφορετικοί φορεί και έχουν διαφορετικό ρόλο, παρόλο που δραστηριοποιούνται βεβαίω στο ίδιο περιβάλλον. Τώρα, ακούσαμε πολλά για τη ρευστότητα κατά μολία με τον όγκο, βραχυπρόθεσμα κατά μολία με τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια. Ποιος αποφασίζει. Αποφασίζει η αγορά. Αν υπάρχει ρευστότητα αυτό είναι υποφελές για όλους. και υπάρχουν αυτοί που θέλουν να προσανατολιστούν μακροπρόθεσμα αλλά και αυτοί με τη ρευστότητα, επί τη βάση της ρευστότητας αποφασίζουν. Ποιος είναι αυτός ο οποίος λοιπόν βάζει, αποφασίζει τη γραμμή που διαχωρίζει το βράχι από το μακροπρόθεσμο. πρόθεσμο. Οι επενδύσεις αυτές γίνονται στις αγορές, ε, υπεραξία προσπαθούν να παράγουν. Είναι θέμα ορισμού λοιπόν, ε, κάπως αυθαίρετου. Βεβαίω υπάρχει ανησυχία στο κοινό, αλλά αυτή η ανησυχία δεν συνάδει με την πραγματικότητα στι χρηματαγορέ. Και όταν ακούω αυτού του βραχυπρόθεσμου κερδοσκόπου που πουλάνε όταν ε, είναι ψηλά η αγορά και αγοράζουν όταν είναι χαμηλά, μπορώ να σα πω από προσωπική πείρα ότι αν, η, ε, αν, γίνεται, αν, αν το κάνετε αυτό συστηματικά θα χρεοκοπήσετε πολύ σύντομα. Όλα αυτά τα προϊόντα αυτό που κάνουν είναι ότι προσφέρουν ρευστότητα στην αγορά. Προστατεύουν κάποια προϊόντα την άλλων. Αυτό το μοντέλο λοιπόν του βράχη πρόθεσμου με το μάκρο πρόθεσμο ε, ή τα διαφορετικά είδη ρευστότητα δεν ισχύει. Θα ήθελα να σας παρακαλώσω να ολοκληρώσετε. Τρία δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε. Σε δευτερόλεπτα γίνονται οι συναλλαγές. Ε, ορισμένες φορές, αλλά μια επιτυχή συναλλαγή που έχει μακροπρόθεσμα χαρακτήρα μπορεί να κρατήσει δύο χρόνια. Είναι κατακλείδη θα έλεγα ότι με τη Βρετανική εμπειρία ο φόρος αυτός πιστεύουμε ότι είναι μια κύρωση ουσιαστικά, μια ζημία, ένα βάρος που ε, επομίζεται η μικρή επιχείρηση και ο καταναλωτής. Ε, στον επόμενο μιλητή θα ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου. Παρακαλώ, σύντομα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ορισμένοι από τους βουλευτές ε, ρώτησαν τι συζητάμε. Συζητάμε αυτόν τον ίδιο φόρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που έχουν υποβληθεί και ξέρετε ότι ο διάβολος συχνά είναι στη λεπτομέρεια. Ε, ξέρουμε ότι ο φόρος αυτός θα οδηγήσει σε συμπληρωματικό εισόδημα και το εισόδημα αυτό θα είναι αποτελεσματικό. Αυτά είναι λοιπόν τα σωστά θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τόσο εισόδημα θα υπάρξει. Δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι η αντίδραση. Και σας το λέω αυτό γιατί εάν ε, φορολογούν δύο πράγματα, η οικονομικά ισότιμα με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν ε, σημαντικές επιπτώσεις. Δηλαδή τελικά το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Και το θέμα με τα παράγωγα είναι ότι θα μπορέσει κανένας να συνδέσει οποιαδήποτε δυνατότητα με τα παράγωγα. Δηλαδή εάν ένα μοντέλο ε, φορολογεί τρία παράγωγα και το άλλο ένα, θα υπάρχει μία μετατόπιση από τη μία μέθοδο στην άλλη, από το ένα είδος στο, στην άλλη. Και γι' αυτό ε, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά με τα έσοδα που μπορούμε να έχουμε από αυτά. Ποια θα είναι η μετατόπιση δραστηριοτήτων, ποια θα είναι τα πρόβλεπτα δεν ξέρουμε ακόμα. Μπορούμε μόνο να τα αναρωτηθούμε βάσει πιας κάποιας πολύ συγκεκριμένης πρότασης. Αυτό είναι το βασικό θέμα που θέλω να το λύσω. Ευχαριστώ κύριο Σβίλαντ. Έχει κάτι να προσθέσει. Εσείς βέβαια είστε στην Κομισιόν, όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα να μας πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, κοιτάξτε καταρχήν. Εγώ ε, άκουσα γενικά τι γίνεται με την ε, με την κατάσταση αυτή σα παρουσίασα τι διάφορε απόψει από τις Γενικές Διευθύνσεις χωρίς να σα παρουσιάσω την άποψη της Κομισιόν τη ίδια. Δεν εργαζόμαστε πάνω σε μια συγκεκριμένη πρόταση γιατί καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι στόχοι της πρότασης. Ας πούμε, θα μπορούσε κανένα να αντιγράψει το STEM duty του Ηνωμένου Βασιλείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα έβλεπε αυτό γιατί αυτός ο φόρος περιορίζεται σε συναλλαγές σε μετοχές εταιριών που είναι ή καταγραμμένες ή έχουν τη βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν κάτι τέτοιο θέλουμε, άλλο είναι αυτό. Αν θέλουμε όμως ένα φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που καλύπτει όλων των συναλλαγές, τότε θα πρέπει να δούμε και το θέμα της ανταγωνικότητας και της μεταφοράς σε άλλα μέρη του κόσμου. Υπάρχει λοιπόν σημαντική διαφορά ανάλογα με την προσέγγιση που θα επιλέξουμε και γι' αυτό καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτό το σημείο. Και αυτό δεν διαφάνει ούτε συζητήσει μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που κυκλοφορούν χωρί να υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή του τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό το φόρο. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση για να ε, διατυπώσουμε κάποια πρόταση. Δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πρώτα σας ευχαριστώ όλους, είναι σαφές. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην απαρχή αυτής της και στο της και θα έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε στο τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας δώσατε τις απόψεις σας σαν αμπρογνώμονες. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κρίνα που θα προεδρεύσει των δύο επομένων σημείων της ημερησίας διάταξης. We're going to start, continue with. We have an exchange of views on. Λοιπόν, έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων πάνω σε μια έκθεση. It's uh, Wolf Klintz, yes. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ο κύριος Κλέιν είναι εισηγητής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σημειώσει συζητήσουμε σήμερα τη οδηγία αυτή, την αναθεώρησή της, μια οδηγία που τέθησε ισχύ το 2003 και αφορά την δημόσια προσφορά των χρεογράφων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το φυλάδιο που τα συνοδεύει τα χρεογράφα αυτά είναι ένα είδος διαβατηρίου και είχε προβληθεί τότε ότι πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ θα εξεταστεί κατά πώς λειτουργεί αυτό το συνεδευτικό ε, έγγραφο και θα δούμε κατά πόσον υπάρχει μια νομική ασφάλεια, κατά πόσον υπάρχουν κάποιες άλλες απαιτήσει και άρα και ε, γραφειογραφικά εμπόδια. Αυτό ήταν ένα τμήμα της ε, ενδεχόμενε πρωτοβουλίε για καλύτερου διαγωνισμού τη Κομισιόν. Πήραμε διάφορες προτάσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά εδώ έχουμε πανεμπόδιση λόγω πολλών διαβουλεύσεων, Σέζαρ κλπ. Το συμπέρασμά μου ποιο είναι. Σε γενικέ γραμμέ συμφωνώ με τι τροπολογίε που προτείνει η Κομισιόν. Είναι τροπολογία συνήθω τεχνική μορφή. Υπάρχουν όμω δύο σημεία στα οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε. Καταρχήν, η λεγόμενη σύνοψη, δηλαδή υπάρχει αυτό το φυλάδιο και έχουμε μετά την σύνοψη που είναι πιο σύντομη, και η Κομισιόν προσπαθεί να τη δώσει μεγαλύτερη αξία σε συνδυασμό και με κάποιες ευθύνες που πρέπει να φέρονται. Κατερχήν, είναι σαφές και εντάξει η Κομισιόν να έχει στόχο ανταγωνιστικά μεταξύ τους προϊόντων, επενδύσεις, ε, χρεόγραφα, ε, ασφαλή ζωής κλπ. να τα καταστήσει όλα αυτά συγκρίσιμα. Ήδη τον Απρίλιο του 2009, δηλαδή πριν από 6 μήνες, προετοίμασε μία ανακοίνωση για τα λεγόμενα PRIPS, που αφορούν τα επενδυτικά προϊόντα για τον μικρό επενδυτή. Είναι καλή αυτή η προσέγγιση, η οποία συστήθηκε και πλησιά, εδώ στην Επιτροπή μας και πάντα ζητάγαμε ακριβώς τα προϊόντα τα οποία ε, προορίζονται για τους μικρούς ε, επενδυτές να υπάρχουν στι ίδιε κανόνες. Τώρα όμω μου φαίνεται ότι εδώ ε, προτρέχουμε τμήματων της νομοθεσίας λείπει δηλαδή ο σαφής προσανατολισμός βιαζόμαστε να εισαγάγουμε μία ιδέα βασικών πληροφοριών χωρίς να έχει οριμάσει η πρόταση και να μην έχει μελετηθεί εις βάθος. Και γι' αυτό δεν είναι σύμφωνη με τον στόχο της καλύτερης διακυβέρνησης. Θα ήταν καλό λοιπόν να περιμένουμε και μετά, όπως προβλέπεται στην αρχή πρίψε, να υπάρχουν οριζόντια ενιαία μέτρα. Αυτό που έχουμε τώρα ίσως υπερβάλλω κάπως, είναι κάπως υπερβολικά ξαφνικό. Και αντί να βοηθήσουμε, έχουμε περισσότερο κατακαιρματισμό. Ο ορισμός δηλαδή των βασικών πληροφοριών, των πληροφοριών κλειδί, θα πρέπει να μελετηθεί καλύτερα. Υπάρχουν κάποια σημεία με τα οποία συμφωνώ. Παραδείγματος ο ορισμός του ε, ικανού επενδυτή όπως τη ΜΥΦΙΤ είναι σωστός. Όσον αφορά την έκδοση ομολόγων ε, και άλλων παρομοίων χρεογράφων θα πρέπει να επιλεγεί η χώρα έκδοσης ακόμα και αν το χρηματιστήριο που τα υπογράφει είναι σε μια άλλη χώρα Εντάξει, αυτά είναι σωστά. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο. Ο καταράχτης λιανικής πώλησης, όπως λέμε. Δηλαδή κάποιο Ινστιτούτο εκδίδει ένα χρόνο, μετά υπάρχει κάποιος ενδιά, με, κάποιος ο οποίος προσφέρει αυτό το χρεόγραφο στην αγορά και αναρωτιόμαστε τώρα ποιος είναι τελικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτού του φυλαδίου. Ο αρχικός εκδότης ή εκείνος που είναι ο τελευταίος μεσάζων που χρησιμοποιεί αυτό το φυλάδιο. Εάν το φυλάδιο αυτό χρησιμοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του πρώτου εκδότη, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι νομικός, αλλά ακριβώ επειδή νομικό ίσω ε, το καταλαβαίνω αυτό το θέμα, θα πρέπει ο πρώτο εκδότη να παραμείνει υπεύθυνο. Εάν δεν υπάρχει όμω η σύμφωνη γνώμη, γιατί κάτι έχει αλλάξει, θα πρέπει εκείνο που το χρησιμοποιεί τελευταίο να φέρει και την ευθύνη. Θα πρέπει επίση να εξετάσουμε την διάρκεια ισχύω του ενημερωτικού αυτού εγγράφου. Η πρώτη Κομισιόν είναι να διευρυνθεί η διάρκεια ισχύω από 12 σε 24 μήνες. Μου φαίνεται λογικό αυτό, γιατί αυτό διευκολύνει τα πράγματα, μειώνει και το κόστος. Είναι σαφές ούτως ή άλλως ότι όταν έχει εισαχθεί κάποιο προϊόν, πρέπει να γίνουν προσαρμογές. Το Συμβούλιο, το οποίο προσπάθησε πριν από το τέλη του έτους να φτάσει σε μια συνεντική άποψη, επανήλθε στους 12 μήνες. Μου φαίνεται περίεργο αυτό. Και όσον αφορά το βασικό ενημερωτικό φυλάδιο, ο εκδότης δηλαδή ε, εκδίδει ένα ενημερωτικό έγγραφο γνωρίζοντας ότι δεν θα εκδώσει τα χρόγραφα αυτά μια φορά αλλά ξανά πάλι μέσα στη διάρκεια 2-3 ετών υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ένα βασικό φυλάδιο το οποίο θα μπορέσει μετά να προσαρμοστεί και πιστεύω ότι αυτό το ο βασικό ενημερωτικό φυλάδιο θα πρέπει να παραταθεί στην ίσχυ του σε 36 μήνες και όχι σε 24. Και το Συμβούλιο εκεί δεν είναι πολύ σίγουρο και πρέπει να το συζητήσουμε το Συμβούλιο. Δύο συμπληρωματικά σημεία. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ θετικό που στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση εκδίδει χρεόγραφα μόνο για τη συμμετοχή στην επιχείρηση των εργαζομένων της επιχείρησης αυτής, θα πρέπει να είναι πιο απλουστευμένες οι απαιτήσει. Αυτό είναι λογικό μου φαίνεται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό και το ίδιο είναι σωστό ότι όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα αναλογικότητας για να απλουστευτεί το θέμα. Όπως είπα και προηγουμένως, το Συμβούλιο προσπαθεί γλίγορα σχετικά να φτάσει σε μια συνένεση. Σήμερα ακριβώς συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών και ίσως έχουν και το θέμα αυτό επιτάπτως και θα προσπαθήσουν με απόφαση πλειοψηφίας να συμφωνήσουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω πολύ τη βιασύνη του Συμβουλίου. Γιατί δεν θα επιταχυνθεί έτσι όλη η διαδικασία. Θα πρέπει εμείς το Κοινοβούλιο να εξετάσουμε το θέμα βάσει του χρονοδιάγραμματός μας και πριν συμφωνήσουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας, δεν μπορούμε να περάσουμε στον τριμερή διάλογο. Φαντάζω ότι οι Σουηδοί έχουν πολύ φιλόδοξο σχέδιο να μπορέσουν μέχρι τα τέλη του να ολοκληρώσουν χι αριθμό φακέλων. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω τη βιασύνη αυτή. Εμείς προβλέπουμε την έκθεση να την υποβάλουμε σε 11 Ιανουαρίου 26-27 να την παρουσιάσουμε μάλλον, 22 Φεβρουαρίου οι τροπολογίες και τέλη Μαρτίου να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Um, e Ο σκέδης ηγητής του ΕΛΚ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η οδηγία έχει δύο βασικούς στόχους. Προστασία των επενδυτών, αποτελεσματικότητα της αγοράς. Οι δύο στόχοι εντάσσονται στην ίδια αρχή, την διαφάνεια. Και υπ' αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξετάσουμε την πρόταση που έχουμε επιτάπητος. Μετά το πακέτο των ε, επενδυτικών προϊόντων ο στόχος δεν είναι πολιτικός, είναι τεχνικός. Νομική ασφάλεια, μείωση του διοικητικού άχθος και αποτελεσματικότητα της αγοράς. Πράγματα ιδιαίτερα ακόμα πιο σημαντικά σε περίοδο κρίσεως. Δεν θα ήθελα να είμαι διεξοδικός, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν θέματα εντελώς ανώδυνα που αφορούν την κοινοτική φιλοσοφία, την νομοθετική εναρμόνιση, τις πληροφορίες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν άλλες προτάσεις που θα πρέπει να βελτιωθούν από τεχνικής νομοθετικής απόψεως, ας πούμε η επιλογή του κράτους προέλευσης, θέμα που και προηγουμένως αναφέρθηκε, και υπάρχουν και άλλα τρίτη κατηγορία θεμάτων που δημιουργούν πολλές ανησυχίες και αμφιβολίες. Το πρώτο αφορά την μη υποχρέωση του ισχύω του προσπέκτους σε περίπτωση επαναπόλυσης. η επαναπόληση είναι ουσιαστικά μια νέα προσφορά. Αλλά αλλάζει η ευθύνη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σχετικά με τον καθορισμό του νομοθετικού καθεστώτος που ισχύει, του φαρμοστού δικαίου, με άλλα λόγια. Θα ήθελα να καταστεί σαφές ότι έτσι πως ε, παρουσιάζεται η περίληψη, το προσπέκτους αυτό, ε, στην ε, πρόταση θα πρέπει να μας κάνει να κατανοήσουμε ότι για ακριβώς αυτό πρόκειται για περίληψη, για σύνοψη όχι για λογοτεχνικό έργο. Συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο κύριος Κλίντς για τις χρονικές προθεσμίες. 36 μήνες είναι νομίζω μια σαφής και θετική πρόταση. Και υπάρχει και η προθεσμία δημοσίευσης τροποποιήσεων. Θα πρέπει να έχει λήξει η διαδικασία προσφοράς. Να έχει δηλαδή ε, παρέλθει το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά. Είναι βεβαίω δύσκολο το έργο εξέβρεση συνένεση, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ πολύ, κύριε Φέιο. Η κυρία Στήλερ. Στέιλερ προφέρεται. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ τον Σκιώδη επίσης ο κύριος Κλίντς έδωσε μια σαφή εικόνα των θεμάτων που μας απασχολούν και όσοι είμαστε καινούργοι μάθαμε πολλά. Τρία στοιχεία που προκέπτουν από τη σημερινή αρχική συζήτηση. Όπως είπε ο εισηγητής και ο σκιώδης ε, εισηγητής από το ΕΛΚ, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα της ευθύνης και ότι το κείμενο θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ενώ η σύνοψη, το προσπέκτους, θα πρέπει να έχει πρακτικό προσανατολισμό και δεν υποκαθιστά το σύνολο των πληροφοριών που θα πρέπει να υπάρχουν. Η χρησιμότητα, ο πρακτικός χαρακτήρας του προσπέκτους είναι το ζητούμενο. Ε, θα πρέπει να το λέμε έτσι απλά, όπως είναι απλά τα αγγλικά, τα δικά μου τουλάχιστον αγγλικά ή σκοτσέζικα όπως το πάρει κανείς. Τέλος πάντων, υπάρχει και το άρθρο 16 που άρει την ευθύνη δημοσίευση στο προσπέκτους κάποιων πληροφοριών και αναφέρει ότι θα πρέπει να είναι ενημερωμένο ανεξάρτητα αν οι ομολογίες υπόκεινται σε, σε ρυθμιζόμενη αγορά ή όχι. Τόσο πάνω είναι πολυτεχνικά αυτά τα στοιχεία. Αλλά το άρθρο 16 θα πρέπει να το δούμε. Για την παράταση της περίοδου ισχύω. Δεν έχω πιστεί. Δεν έχω πιστεί. 12 ε, μήνες είναι η ισχύουσα προθεσμία. Προτείνεται τώρα να πάει σε 24. Η ανησυχία μου είναι ότι οι επενδυτές να έχουν στα χέρια τους στην αρχή της περίοδου ένα προσπέκτους με κάποιες πληροφορίες και μετά τους 24, 12, 24 όσοι είναι μήνες να λάβουν ένα δεύτερο διαφορετικό και άρα να προκληθεί κάποια σύγχυση. Δεν είμαι πεισμένη λοιπόν για τον πρακτικό χαρακτήρα αυτού του μέτρου. Επανέρχομαι ε, στη σύνοψη και το PRIPS. Είναι σημαντική η συνέπεια μεταξύ των νομοθετημάτων. Και ο κύριος Κλίντς έχει απόλυτο δίκιο που θέτει θέμα συνέπειας με το ΠΡΙΠΣ. Ευχαριστώ. Μας δώσατε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για πρώτη φορά αυτό το θέμα. Είναι κρίμα που είμαστε ε, ολιγάριθμοι, αλλά εντάξει, τεχνικό είναι το ζήτημα, δεν δημιουργεί και πάθη. Η κυρία Γκέρι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις σκέψεις που εξέφρασε. Όλα αυτά που μας είπε τα βρίσκω πολύτιμα και έχω δύο παρατηρήσεις. Όσον αφορά την σύνοψη και την πληροφόρηση, ο κύριος Κλίντς επισήμανε ήδη ότι στην πρόταση της Κομισιόν δεν είναι απόλυτα σαφέ το θέμα της ενημέρωσης. Πρέπει λοιπόν να το διευκρινίσουμε, να πούμε τι θα είναι ενημέρωση και τι θα είναι ανακεφαλαίωση. Είναι λοιπόν σημαντικό η περίληψη ανακεφαλαίωση να μην ε, διατυπώνεται με τεχνικά λόγια, αλλά με πολύ πιο κατανοητά, απλά. Κάτι άλλο. Ε, σχετικά με αυτό το έγγραφο, το ενημερωτικό δελτίο και με την ε, αστική ευθύνη. Ποιος φέρει δηλαδή την ευθύνη. Η πρόταση της Κομισιόν έχει ως στόχο να επεκτείνει την αστική ευθύνη σε όλα. Παραδείγματο χάρη, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση, μία απόφαση που δεν είναι τεκμηριωμένη, γιατί οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό αυτό τεύχος ε, δεν είναι επαρκείς, τότε θα ήταν σωστό η αστική ευθύνη να αφορά κάθε πρόταση που περιλαμβάνεται στο τεύχος. Και νομίζω αυτό προστατεύει τους επενδυτές εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο. Ο εισηγητής λοιπόν έχει το λόγο, ο κύριος ε, Κλίντς. Ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους για τις ε, παρατηρήσεις τους. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος όπως ο συνάδελφος κύριος Φέο από την ε, Πορτογαλία που λέει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ε, συμβιβασμό. Αν δεν το λέω καλά, δεν σα κατάλαβα καλά. Ε, νομίζω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο θα επιτύχουμε τελικά το συμβιβασμό. Τώρα, κατά πόσον στην τριμερή συνάντηση με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, κατά πόσον εκεί θα συμφωνήσουμε, θα δείξει. Νομίζω ότι σε τελική ανάλυση, επειδή τώρα πια έχουμε και μεγαλύτερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη ισχύ δεν πρέπει να παραιτηθούμε τόσο εύκολα. Αυτά που αναφέρθηκαν είναι θέματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε ε, και εγώ βέβαια θα τα εξετάσω Πάντω, ε, καλό είναι καταρχήν να συμφωνήσουμε για το στόχο. Δηλαδή, στόχος είναι να βελτιώσουμε την κοινή αγορά, να βελτιώσουμε την προστασία του επενδυτή και σίγουρα θέλουμε λιγότερη και όχι περισσότερη γραφειοκρατία. Νομίζω λοιπόν ότι όσον αφορά αυτούς ε, τους ε, στόχους πράγματι ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε στο εγχείρημα που έχουμε αναλάβει να επιφέρουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. 26 Ιανουαρίου θα εξεταστεί το σχέδιο της έκθεσης 22 Φεβρουαρίου, καταληκτική μερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών και κατόπιν εξέταση των τροπολογιών 16 και 17 Μαρτίου. Τώρα λοιπόν πάμε στο σημείο υπαριθμών 18 της ημερήσιας διάταξης. Η συγητής εδώ είναι ο κύριος Κάζα. Πρόκειται για την έκθεση προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφή τη επιβάρυνση για τι παραδόσει ορισμένων αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που είναι πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο απάτη. Ευχαριστώ. Με μένα αρχίσαμε τη συνεδρίαση αυτή, με μένα τελειώνουμε. To, to combat... Σύμπτωση. Λοιπόν, καταπολέμηση του ΦΠΑ, ε, πάτη καρουσέλ κτλ. Ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι, ομιλώ. Οι απάτες του ΦΠΑ ανησυχούν όλα τα κράτη-μέλη διότι ε, αφορούν την ορθή λειτουργία της ιστορικής αγοράς αλλά και την συλλογή εισοδήματος. Ο missing trader είναι εδώ το ε, θέμα μας. Αυτό του είδους η απάτη οργανώνεται με ευκόλως μεταφερόμενα προϊόντα με υψηλή αξία όμως εξαπλώνεται και στον τομέα των υπηρεσιών και αυτό που μας ανησυχεί είναι η ανίχνευση ε, ε, των απατών που αφορούν την ανταλλαγή των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος από business to business καταβάλλεται ο ΦΠΑ και όχι από την επιχείρηση στο κράτος μετά ζητείτε επιστροφή του ΦΠΑ και έτσι ο τελικός καταναλωτής είναι αυτός που φέρει το που ζημιώνεται διότι ως φυσικό και μη νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ. Αλλά το B2B στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το ισχύον σύστημα ΦΠΑ δεν χρεώνει ΦΠΑ από τον πάροχο. Άρα τα αγαθά αυτά κυκλοφορούν χωρίς ΦΠΑ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Η απάτη λαμβάνει η χώρα όταν ο παροχός χρεώνει και παίρνει το ΦΠΑ από το πελάτη του σε ενδοκινοτική συναλλαγή και μετά επιστρέφεται το ΦΠΑ από το κράτος χωρίς όμως να τον έχει καταβάλει ο α, έμπορος. και έτσι για ένα μόνο προϊόν ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα πολλές φορές. Εξού και όρος καρουσέλ. Στον Ηνωμένο Βασίλειο οι απάτες αυτές γαϊτανάκι είναι 24% του συνόλου των απατών του ΦΠΑ. Και βεβαίως δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό η Κομισιόν δημοσίευσε μία μελέτη σύμφωνα με την οποία το ποσό μπορεί να φτάσει στην περίοδο 2000-2006 μέχρι 139 δις ευρώ. Στα πλαίσια του συστήματος ανταλλαγών εκπομπών διοξιδίων του άνθρακου, το άνθρακος, οι συναλλαγές αυτές γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό αυτή η συναλλαγή φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του εμπορευομένου. Αγοράζει κάποιες μονάδες ε, ο ενδιαφερόμενος που τις πουλάει μετά σε επιχειρήσεις κρατών μελών με το ΦΠΑ που εκεί ισχύει. Δεν καταβάλει το ΦΠΑ όμως το κράτος μέλος από τον έμπορο και οι περισσότερες ε, ανταλλαγές ε, θα έγιναν το 2003. Είναι κάτι το οποίο έπληξε την αξιοπιστία του συστήματος και γι' αυτό η Κομισιόν θέλει να, να λάβει άμεση δράση για να επιδιορθώσει την ε, κατάσταση για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστεί η αντιστροφή ε, του βάρους, της απόδειξης. 5 με 10% των επιδοτήσεων αυτών ε, γίνονται δυνάμει του συστήματος του Κιώτο με δημοπρασίες από με, σύν το χρόνο ε, οι, όλες σχεδόν οι συναλλαγές θα γίνουν έτσι. Μέχρι τώρα υπάρχουν διάφορα άλλα μέσα, ιδιωτικά, δηλαδή μεταξύ των εμπορευμένων σε μια επιχείρηση και σε διάφο... διασυνοριακά, διαμεθοριακά δεύτερον με τη μεσολάβηση ενό διαμεσολαβητή και τρίτο spot market ε, σε μια από τις αγορές της ε, Ευρώπης για την κλιματική μεταβολή. Η πρόταση δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014 και για μια ελάχιστη διετή περίοδο να εισαγάγουν και να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό της αντιστροφής για έναν προκαθορισμένο κατάλογο υπηρεσιών και προϊόντων. Αυτός ο μηχανισμός θα δώσει τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις που έχουν ΦΠΑ να πουλούν αυτά τα προϊόντα σε άλλη επιχείρηση χωρίς ΦΠΑ. Ο φόρος ε, συλλέγεται μόνον όταν πωλείται το προϊόν ε, σε επιχείρηση που δεν έχει ΦΠΑ ή σε ιδιώτη. Αυτός είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή διότι δεν έχει ποτέ καταβάλει ΦΠΑ. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα για απάτη καρουσέλ. Γαϊτανάκι. τρία πρέπει να είναι τα αντικείμενα της συναλλαγής με maximum δύο προϊόντα και μία υπηρεσία. Και υπάρχουν και υποχρεώσεις όπως ο, υποχρέωση για οποια, ανακοίνωση του ονόματος οποιοδήποτε φορολογούμενου προσώπου, πρόληψη ε, απατών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ε, της εφαρμογής του συστήματος. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εν λόγω μέτρα και πρέπει να το κάνουν ε, σύμφωνα με τη συνολική αποτελεσματικότητα ε, του συστήματος. Υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν, παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Πρώτον, τροπολογία υπερθμών 5 θα πρέπει να καταστεί σαφέστερο ότι η εφαρμογή του προαιρετικού μηχανισμού αντίστροφης του βαρουσιαπόδειξης αφορά μόνο του, τις ε, ε, που υπάγονται σε αυτό το μηχανισμό. Αν αποφασίσει ένα κράτος μέλος να χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή, η αντιστροφή θα πρέπει να είναι δυνατή και στα πλαίσια της ανταλλαγής του εμπορίου των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος εξού και οι τροπολογίες 2 και 6 που λένε ότι όταν ένα κράτος μέλος επιλέξει να εφαρμόσει αυτό το σύστημα θα πρέπει να περιλάβει πιστοποιητικά εμπορίας ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος γιατί ένα μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει την περίπτωση ε, απώλειας εισοδήματος όταν το ποσό της απάτης είναι υψηλότερο από το εισόδημα. Υπάρχει αβεβαιότητα για το πόσο ο μηχανισμός θα επηρεάσει άλλους τομείς του εμπορίου ή θα μετατοπίσει το κέντρο βάρους της απάτης προς άλλα κράτη-μέλη. Οι τροπολογίες 7 και 8 για τις υποχρεώσει των φορολογουμένων και τη μείωση, την ελαχιστοποίηση του διοικητικού άχθους και τη γραφειοκρατία για τι επιχειρήσει. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα είτε να ζητούν εκθέσεις ανασυναλλαγή είτε μία έκθεση για όλες τις συναλλαγές. Η τροπολογία 9 έχει λόγους συγκρισιμότητος που θα πρέπει να από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ προτείνω η Επιτροπή ΦΠΑ να διαβουλεύεται με τα κράτη-μέλη, μάλλον να ζητούν τη γνώμη της στα κράτη-μέλη πριν αποφανθούν για την αποτελεσματικότητα του συστήματος και τις ενδυνάμει συνεπιές του για τις απάτες. Οι τροπολογίες 4 και 10. Αναφέρω εδώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερωθούν για την συνολική αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της αντιστροφής του βάρους απόδειξης και για όλες τις ενδεχόμενες προτάσεις που ενδεχομένως να υποβάλει στο μέλλον η Κομισιόν, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την αποτελεσματικότητα τη εφαρμογή του συστήματο αυτού μέχρι τον Ιούλιο του 2014. Μέσω αυτών των προτάσεων η πρόθεσή μου είναι να ενδραμώσουμε την ασφάλεια και την αξιοπιστία του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών ενώ συγχρόνως να μειώσουμε το διοικητικό άχθος για τις έντιμες επιχειρήσεις. Ε, είμαι πεπισμένο. ε, να διασφαλίσουμε επίση ότι θα ενημερωθεί πλήρω το Κοινοβούλιο εις ό,τι αφορά ενδεχόμενε μελλοντικέ προτάσεις με το ίδιο θέμα Αυτά, ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάζα Α, ο κύριος Βίνξεν ε, ναι, εδώ, εδώ, εδώ Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε και θέλω να σας πω χαίρομαι που ε, καθιστά την οδηγία σαφέστερη και παράλληλα μειώνεται ο κίνδυνος απάτης στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να υποβάλω. Πρώτον, όσον αφορά το παράρτημα εδώ αναφέρεται με σαφήνεια ποια μορφή θα πρέπει να λάβει αυτός ο κατάλογος. Και προφανώς ε, ο κατάλογος αυτός ε, αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι ε, στην οδηγία θα συμπεριληφθούν και αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν όμως όλες τις χώρες. Να μπορεί δηλαδή ο κατάλογος να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις και να ορίσουν και κριτήρια αξιολόγησης. Όμως αυτά κριτήρια μπορεί να ποικίλουν στα κράτη-μέλη. Και ερωτώ ε, κατά πόσον... Ε, γνωρίζετε ότι το αποτέλεσμα θα είναι δύσκολο να συγκριθεί και μετά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να αξιολογήσει κανείς το σύστημα. Ε, δεν θα μπορεί κανείς να πει κατά πόσον η εφαρμογή του συστήματος ήταν επιτυχής ή όχι. Ο εισηγητής κατέθεσε μια τροπολογία, δεν υπαριθμών 10, όπου αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή των υπαριθμων 10 οπου αναφερεται πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σχετική έκθεση. Ε, διερωτώ λοιπόν κατά πόσον μπορούμε να διευκρινίσουμε λιγάκι την ε, οδηγία προβαίνοντα σε αξιολόγηση των επιπτώσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο κατά πόσον θα πρέπει το σύστημα αυτό να ε, εφαρμόζεται εσαΐ ή όχι. Αναφέρουμε πάντα σε υπηρεσίες, αγαθά που μπορούν να καταστούν αντικείμενο απάτης. Και τέλος ε, να πω ότι ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λούτριξεν, ο κύριος Βολφ Κλίντς δεν έχω πολλά να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κάζα για τη δουλειά του. Όσον αφορά το θέμα της απάτης στον ΦΠΑ, το θέμα αυτό υπάρχει στη μερίσια διάταξη εδώ και χρόνια. Και αν ακούσει κανείς τα στοιχεία, κανείς δεν τα γνωρίζει επακριβώς. Περίπου τα λέει κατά προσέγγιση, τα υπολογίζει. Και γι' αυτό γίνεται κατανοητό πόσο καιρό χρειάζεται έτσι ώστε να περιοριστούν τουλάχιστον αυτές οι απάτες. Γιατί εδώ ε, πρόκειται για δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει λοιπόν να επέλθει κάποια τάξη και ελπίζω ότι θα συνεργαστούν τουλάχιστον αρκετά κράτη-μέλη. Ίσως να μην κατάλαβα καλά, αλλά εξακολουθώ ε, να πιστεύω ότι ε, τελικά αυτό το σύστημα δεν θα το εφαρμόσουν όλα τα κρατημέλη παρά μόνο κάποια από αυτά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η προσπάθεια αυτή να επιτύχει γιατί αν αποτύχει ε, θα είμαστε πάλι στο σημείο μηδέν εκεί που ήμασταν πριν από 20 χρόνια. Θα κλεγόμαστε όλοι και τίποτα δεν θα γίνεται. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταστεί δυνατόν να υπάρξει αντιστροφή της επιβάρυνσης και τελικά αυτή η δήλωση περί ΦΠΑ αποτελεί απλούστευση γιατί κατά κάποιον τρόπο όλη αυτή η αλυσίδα συρρυκνώνεται σε ένα και μόνο άτομο. Όμως, και εδώ έρχεται όμως, όμως φοβάμαι ότι και με αυτή την προσέγγιση δεν θα μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν απάτες. Οι εγκληματίες είναι ιδιαίτερα δημιουργικοί, ε, έχουν φαντασία και εδώ λοιπόν θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που υπάρχει μια επιχείρηση η οποία είναι η τελευταία στην αλυσίδα και δέχεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, αγοράζει αυτό και πρέπει να αποδώσει τον ΦΠΑ, παράλληλα όμως αυτή η επιχείρηση ε, δέχεται και επιστροφή ΦΠΑ γιατί απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Ε, τελικά αυτή η επιχείρηση μπαίνει σε αυτό το σύστημα ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσει το προϊόν, απλά το μεταβάζει περαιτέρω. Παρ' όλα αυτά υποχρεούται σε δήλωση ΦΠΑ, ε, δέχεται επιστροφή του ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Οφείλουμε λοιπόν να προσέξουμε έτσι ώστε από το παράθυρο να μην ε, προκαλέσουμε επιπρόσθετο διοικητικό ε, κόστος. Γιατί κατ' ουσίαν ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να είναι και σίγουρος ότι ο αποδέκτης ε, τα κάνει όλα σωστά. ΦΠΑ, αφημί, πρόκειται δηλαδή για ένα γραφειοκρατικό έλεγχο που όμως πρέπει να γίνει σωστά. Αλλιώς ε, ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες ε, στην απάτη και στην περίπτωση του πάροχου υπηρεσιών ε, προκύπτει και διοικητικό άχθος, ε, άρα δηλαδή πρέπει κάπως να τα συγκρατήσουμε όλα αυτά. Τίθεται και το εξής ερώτημα. Σε τελική ανάλυση, αν παρόλα αυτά εμφανιστούν περιπτώσεις απάτης, ποιος ευθύνεται, ποιος φέρει την αστική ευθύνη του ο πάροχος της υπηρεσίας ή μήπως ο αποδέκτης ή κάποιος άλλος. Εγώ προσωπικά έχω πολύ περιορισμένο αριθμό τροπολογιών, 5-6 είναι που νομίζω ότι θα βοηθήσουν στη διευκρίνηση των απόψεων του εισηγητή. Θα τα βρούμε πολύ γρήγορα στο ποια πρέπει να είναι η τελική διατύπωση και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε με την Επιτροπή, ούτε με το Συμβούλιο και αυτή μας η προσπάθεια θα εμποδοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκιούρη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κάζα για αυτή την ε, θαυμάσια ε, έκθεσή του και το πολύ ε, ικανοποιητικό υλικό που συνέλεξε ένα πολύ δύσκολο θέμα που μας το παρουσίασε με θαυμάσιο τρόπο. Έχω δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Εργαζόμαστε, σήμερα το πρωί μάλλον, μιλήσαμε ήδη για την φοροδιαφυγή και εγώ είπα ότι οι δικοί μου οι συμπολίτε είναι ιδιαίτερα εφάνταστοι στον τομέα της φορολογικής απάτης. Το ίδιο ισχύει και για την απάτη γαϊτανάκη, όπως αποκαλείται. Έχω μία ερώτηση. Δίνουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα επιλογής. Μπορούν να επιλέξουν ε, σε ποια τρία θέματα θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης. Εγώ όμως ήθελα να διευρύνω ε, τον κατάλογο και για τα προϊόντα της πληροφορικής. Ακριβώς διότι στην Ουγγαρία έχουμε πολλές καταχρήσεις με προϊόντα πληροφορικής. Ε, θα ήθελα λοιπόν να διευρύνω τον κατάλογο συμπεριλαμβάνοντας και αυτά τα προϊόντα. Και άλλη μία παρατήρηση. Ο κύριος Κλίντς είπε ότι δεν πρέπει να ε, διευρυνθεί, να αυξηθεί το διοικητικό άχθος. Ότι πρέπει να το συρρυκνώσουμε, μάλιστα. Και ρωτώ τον εισηγητή. Αν ορίζαμε ένα κατώτατο όριο, κάτω από το οποίο δεν θα πρέπει να εισάγουμε αυτό τον ε, μηχανισμό αντιστροφής ε, της ε, επιβάρυνσης. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν σωστό. Αν είμαι σωστά ενημερωμένη, ίσως να κάνω λάθο, λάθος, στη Γερμανία αναφέρεται ένα τέτοιο κατώτατο όριο της τάξης των 5.000 ευρώ. Εσείς τι λέτε γι' αυτό κύριε Σιγητά. Τέμπιτ, θέλετε να απαντήσετε. Κοιτάξτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εσκαιώδεις με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Η πρώτη εκδοχή του εκδοσίας μου. Ε, ναι, μιλάμε για απάτη και όσο και αν προσπαθήσουμε, η απάτη δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Πολλά χρόνια συζητάμε το θέμα της απάτης όπως δικαίως ε, παρατήρησε ο κύριος Κλίντς. Και δεν πρόκειται να εξαλείψουμε πανελώς την απάτη θα πρέπει μόνο να περιορίσουμε τις δυνατότητες για απάτη. Υποβλήθη μία, μία σειρά ε, ιδεών από τους συναδέλφους με τους οποίους μπορώ να συμφωνήσω. Τώρα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι περαιτέρω τροπολογίες που θα μπορούσαν να υποβληθούν για να είμαστε σίγουροι. ότι αυτό που κάνουμε δεν θα αποτελέσει συμπραγματικό άχθος για τις επιχειρήσεις μας. Ούτε διοικητικό άχθος, ούτε οικονομικό. Και όσον αφορά την πρόταση για τα κατόφλια, ξέρω ότι στο Ρωμανό Βασιλείο υπάρχει ένα κατόφλι και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε ίσως να λάβουμε υπόψη. Η αξιολόγηση του σχεδίου αυτού πιλότου που είναι εθελοντικό για όλα τα κράτη-μέλη θα οδηγήσει σε μια αξιολόγηση από την Κομισιόν γιατί τότε θα δούμε πώς λειτουργούν τα σχέδια αυτά και μετά θα υπάρχει μια τελική αξιολόγηση πριν εισαχθούν οι μηχανισμοί μόνιμα. Το, στο Κοινοβούλιο ζητάμε λοιπόν να παραμείνουμε ενήμεροι, να ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα που θα έχουν καταγραφεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός και πρέπει να φροντίσουμε το σύστημα και ο μηχανισμός να είναι φιλικό κατά το δυνατόν προς τις επιχειρήσεις. Εγώ συνάντησα εκπροσώπους του τομέα και τα προβλήματα που οδήγησαν εδώ μου είχαν ήδη αναφερθεί προηγουμένως. Θα πρέπει τώρα να συζητήσουμε με το Συμβούλιο, με την Κομισιόν, με τον επιχειρησιακό κλάδο, που προφανώς θα πρέπει να προστατευτεί από αρνητικές επιπτώσεις που θα προέρχονται από την πρόταση αυτή. Ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Is it working now? The, uh, the 8th of December is the deadline for amendments. Λοιπόν, υπάρχει προθεσμία για στεροπολογίες. 11 Ιανουαρίου θα τις εξετάσουμε και η ψηφοφορία θα γίνει 27 Ιανουαρίου 2010. Well, this brings us to the... Εδώ τελειώνουμε τις εργασίες μας. Η μνήμη της επόμενης συνεδρίασης είναι την επόμενη Δευτέρα, 7 το μηνός, στις 2 το μεσημέρι, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.